Ok. Chers collègues, bonjour. Je sais, je vous ai manqué pendant un quart d'heure. Ξέρω ότι σας έλειψα για ένα τέταρτο καλημέρα σας, αλλά κατέφθασα. Δεν ξύπνησα αργά. Είχα πρόγευμα με κάποιον, κάποιαν. Déjeuner de travail. Πρόγευμα εργασίας. Monsieur, Marinescu, vous êtes Κύριε Μαρινέσκου, εσείς ήρθατε στην ώρα σας. Ωραία. Ας αρχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Λοιπόν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές κατά τη χτεσινή συνεδρίαση βλέπετε τα πρακτικά. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι τις 12.30 τότε θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα δούμε κατά πόσο έχουμε επαρκή αριθμό. Άρχεται η ψηφοφορία για να δούμε αν έχουμε απαρτία, δοκιμή, πέρας. Ωραία, όλα έχουν καλός. Αρχίζουμε λοιπόν καταρχήν απαλλαγή 2016 της Επιτροπής. Δεμόντε. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 12 άρχεται πέρας απορρίπτεται όμικρον α1. Στην προφορική, προφορική Μαρινέσκου, υπέρ. Καταρχήν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική. Α, είσαστε τυχερός κύριε Μαρινέσκου, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο ηλεκτρονικά. Πέρας. Υπέρ 37. Τέσσερις κατά. Κυρία Ντεμόντε, εγκρίνεται η έκθεσή σας και συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε με την έκθεση Φέρμπερ για τους σιδηροδρόμους. Καλημέρα σας κύριε Φέρμπερ. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές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 Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Φέρμπερ. Ωραία συνεχίζουμε. to Δική σας έκθεση κύριε Φέρπερ. 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Κύριε Νταλούντε, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεσή σας. Συνεχίζουμε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη θαλάσσια ασφάλεια. Η κυρία Μέσνερ είναι η, η συγγήτρια. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Μάισνερ. Εγκρίνεται η έκθεσή σας με μεγάλη πλειοψηφία. Σέζαρ. Αρχίζουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ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 Λοιπόν, τώρα περνάμε στη δική μου έκθεση για τις στατιστικές για τους σιδηροδρόμους. Έχουμε μία ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ, ένας κατά. Δεν θα ψάξω αυτόν που καταψήφισε. Ωραία, συνεχίζουμε. Και περνάμε λοιπόν στην επόμενη έκθεση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Συνεργατικά και Εφηγή Συστήματα Μεταφορών. Έκθεση Ουλελή. Ξεκινάμε. 33. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Άποχες. γιατί 35. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 51. Πέρας. Απορρίπτεται η 51. 55. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 57. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 70. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Σοσιαλιστές, παρακαλώ, δεν βλέπω πώς ψηφίζετε. Είσαστε υπέρ, μάλιστα. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Λείπε 4. Πέρας. Εγκρίνεται. Λίμπε 2, δεύτερο μέρος παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 7, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. για 19 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Ένδυ 15 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. εγκρίνεται 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 140. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 170 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δύσκολο. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Ηλεκτρονική παρακαλώ, επαλήθευση για την 170. Πέρα. Εγκρίνεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. Μάλιστα. Επαλήθευση αφού θέλετε για την 173. Παρακαλώ, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, απορρίφθηκε. NV25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίπε α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Περνάμε τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. άποχε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και η τροπολογία 10 και τώρα το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Je ferme le vote. 39. Πέρασα τη ε, ψηφοφορία με μεγάλη ε, πλειοψηφία, 39 ψήφοι υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες και συνεχίζουμε με τις εργασίες μας. On peut, après deux minutes, on peut vider les salles, directement commencer à... Je vais demander à ceux qui quittent la... Παρακαλώ, όσοι θέλουν να φύγουν από την αίθουσα, να φύγουν ησύχως. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε παρακαλώ τις εργασίες μας. Όσοι θέλουν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων, παρακαλώ εκτός αιθούσης. Να περάσουμε στην ε, ακρόαση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών συνδρομικών γραμμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόασή μας ε η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εργασιών μας σε ό,τι αφορά την πρόταση αναθεώρηση του κανονισμού 1611 σε ό,τι αφορά τις ε, υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιβατών συνδεδρομικών γραμμών. Ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας πριν από το θερινό διάλειμμα. Και ο σκοπός της ε, ακρόασης αυτής είναι να ακούσουμε τις ε, τοποθετήσεις διαφορετικών εμπλεκομένων φορέων στον θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τους επιβάτες, ε, τις δομικές επιχειρήσεις και εταιρείε και τους ρυθμιστικές αρχές. Ε, προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση όμως και προτού προβούμε στην έναρξη των εργασιών μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπορεογνώμονες οι οποίοι δέχτηκαν να έλθουν και να μας μιλήσουν εδώ ενώπιον της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήλθατε εδώ και που μας ε, τιμάται με την εμπειρογνωμοσύνη σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Οι εργασίες και τα δικαιώματα των επιβατών συνδρομικών γραμμών είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πιο πολλών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω τον ε, λόγο στον ε, εισηγητή, τον κύριο Αντιπρόεδρο Μπόγκουσλαβ Λιμπεράτσκι. Θα έχετε πέντε λεπτά, κύριε Σιγητά, για να κάνετε κάποια προκαταρτικά σχόλια για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πέντε λεπτά σύντομα να μας παρουσιάσει την πρότασή της και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας. Κυρίες και κύριοι, θα έχετε έξι λεπτά έκαστος για να τοποθετηθείτε από πλευρά τη οργάνωσης την οποία αντιπροσωπεύετε και θα τηρήσω αυτή το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια συζήτηση στη συνέχεια μετά τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Σλεύσκη από τις πολιτικές τηλεδρομικές γραμμές ε, που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε από τη Γαλλική Ομοσπονδία ε, Μεταφορών. Ε, να σας καλωσορίσω και εσάς, ε, κύριε Γκαζό. Έχετε πολλή δουλειά στην παρούσα φάση, έτσι δεν είναι. Την κυρία Άντα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηρίας. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας και εσείς τον κύριο Βίλι Σμιόλτερς, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επίβατων. Καλώς ορίσατε και εσείς και καλημέρα σας. Τον κύριο Ρέφν, ο οποίος είναι σύμβουλος της Δανέζικες ε, ε, Συνδρομικές Γραμμές. Τον κύριο Σμιθ, blogger στο blog SIF61. Καλημέρα και σε εσάς, καλώς ορίσατε και τον κύριο Λόχμαν, εκτελεστικό διευθυντή της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Συρρώμων και Υποδομών. ΣΕΡ, CER. Θα γνωρίζουμε καλά. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Σαν να μιλάτε πολύ όμως σήμερα. Και κάνετε φασαρία. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στον εισήγητή μας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και μετά θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο την επωνομαζόμενη ping-pong για να ακούσουμε ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή και στους Κιώδης και στον κύριο Ντένις Ντεγιόγκ, ο οποίος είναι εισηγητής της γνωμοδότησης από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Πού είναι ο κύριος όμως? δεν έχει ακόμα καταφτάσει. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω πολωνικά. Ωραία. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, που ε, κατέστησαν δυνατή αυτή την ακρόαση. Δεύτερον, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη που πρέπει να αποχωρήσω πριν τις 11. Ε, είναι όμως η εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να προεδρεύσω σε συνεδρίαση με εκπροσώπους όλων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων συνάδελφος Ερτούκ θα με αντικαταστήσει και θα συνοψίσει την ε, συζήτηση. Δισεκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν ε, τις σιδηροδρομικές ε, υπηρεσίες κάθε χρόνο και πολλοί από αυτούς ταξιδεύουν πολλές φορές την εβδομάδα, το οποίο σημαίνει ότι οι σιδηρόδρομοι παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες και παράγουν τις υπηρεσίες αυτές. Θα θέλαμε λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των επιβατών στις σιδηροδρομικές μεταφορές Ε, με τις προσδοκίες των επιβατών όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών. Θέλουμε ε, ενοποίηση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλουμε ένας επιβάτης που επιβαίνει σε ένα τρένο στη Βαρσοβία και κατεβαίνει από το τρένο στην ε, Βουδαπέστη που ταξιδεύει μέσω της Πολωνίας, Τσεχίας και φτάνει στην Ουγγαρία να πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζει διαφορετική νομοθεσία. Θέλουμε λοιπόν να ενοποιήσουμε το σύστημα δικαιωμάτων των επιβατών. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε και επιπλέον δαπάνες για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Θέλουμε λοιπόν ποιότητα αλλά σε καλή τιμή. Οι εταιρείε μεταφορών θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν τις ποιοτικέ αυτές υπηρεσίες χωρίς να απειλείται η οικονομική του ε, κατάσταση και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο συμβασμό και κατά τη σημερινή ακρόαση θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις, δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Η πρόεδρός μας ήδη παρουσίασε τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους ε, των επιχειρήσεων, των χρηστών, των ε, ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων με αναπηρίες. Ε, των ε, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ε, τον κύριο Λόχμαν για παράδειγμα. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω όλες τις συνεισφορές σας στην έκθεση που θα πρέπει σύντομα να εκπονήσω. Μπορώ επίσης να σας ενημερώσω ότι είχα τη χαρά να συναντήσω δεκάδες εκπροσώπους από διάφορους οργανισμούς όπως αυτού ε, που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα θα διευρύνουμε τις γνώσεις μας και αυτό θα μας βοηθήσει να διατυπώσουμε και τι τροπολογίες μας και να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, διότι θέλω να τονίσω ότι θέλουμε περισσότερους επιβάτες σιδηροδρόμων και λιγότερους σε άλλα μέσα μεταφοράς σε σωστή τιμή όμως και με τρόπο που να μην απειλούνται τα οικονομικά συμφέροντα των, των σιδηροδρόμων μας. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση λοιπόν με τους εμπειρογνώμονες μας. Να ξεκινήσουμε με τους εκπροσώπους ε, των πολωνικών σιδηροδρόμων. Τον κύριο Λζέσκι, πού είστε. Α, να δώσουμε ίσω πρώτο το λόγο στην ε, πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν σα είδα, αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, μην ξεκινήσουμε με συγκρούσεις. Πρωί-πρωί. Να σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσετε τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Dear uh, Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι για τη σύγχυση. Πολύ σύντομα. Γιατί υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης. Είχαμε μια έκθεση το 2013 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού για τα δικαιώματα των ε, επιβατών των σιδηροδρόμων ε, που έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Έχουμε κατακαιρματισμό στον τομέα αυτών διότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διάφορες παρεκκλήσεις. Δεύτερον, Έχουμε και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές για τα δικαιώματα των ε, ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, κατά την εφαρμογή διαπιστώσαμε ότι κάποιοι όροι και ορισμοί δεν είναι πολύ σαφείς και όσον αφορά τα ενιαία εισιτήρια, τα through tickets. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην πρόταση αυτή δεν μιλάμε για τη δημιουργία του όρου του ενιαίου εισιτηρίου, αλλά απλά αναφέρουμε τις περιπτώσεις όπου ο επιβάτης αγοράζει τέτοιο εισιτήριο ή όχι. Κατόπιν όσον αφορά την ε, εφαρμογή ε, και την ανωτέρα δύναμη, την ανωτέρα βία θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις ε, διότι το δικαστήριο έλεγε ότι δεν μπορούν να ε, εξαιρεθούν από την ε, καταβολή αποζημίωση σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Γι' αυτό θέλουμε να αναδιατυπώσουμε τον κανονισμό αυτόν. Τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε η σχετική δουλειά και θέλουμε από τη μία να έχουμε καλύτερη προστασία των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα και την κατάσταση του τομέα των σιδηροδρόμων. Όσον αφορά λοιπόν το πεδίο εφαρμογή, ε, θέλουμε να ε, αφαιρέσουμε τι παρεκκλήσει. Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίε, θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε πληροφορίε ε, και σε μηχανισμού προσφυγή. Θέλουμε επίση να βελτιώσουμε την παροχή πληροφοριών προ όλου του επιβατέ. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των ενιαίων τερίων και των ε, σχετικών υποχρεώσεων. Και θέλουμε επίσης ε, να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των, ε, του χειρισμού των προσφυγών από τις Εθνικές Συνδρομικές Αρχές και επίσης ε, το θέμα του, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ε, θα πρέπει ε, να μην φέρνουν μόνο συνδρομικές επιχειρήσεις το βάρος αυτό. Θα πρέπει να το πειράζονται με τους διαχειριστές των σταθμών και των υποδομών. Επίσης, σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να έχουμε σχετικές διατάξεις ε, για να αποφύγουμε καταστροφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είχα να πω εν συντομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανημέρωση αυτή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνωμονές μας και στράφουμε λοιπόν πάλι προς εσάς προς τον κύριο Ολσέσκι, εκπρόσωπος είσαστε των ε, πολωνικών συνδρόμων και σας δίνω το λόγο λοιπόν παρά αυτά για έξι λεπτά. Ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την δυνατότητα να πάρω το λόγο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας την πρόσκληση που απευθύνατε στους ε, πολωνικούς κρατικούς σιδηροδρόμους PKP. Οι τροποποίησεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα αποτελέσουν ε, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στον συνδρομικό τομέα στους επόμενους μήνες. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι τεράστιος. Ο κανονισμός 1371 ε, κάθετος 2007 που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των επιβατών εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Και η πολωνικοί σιδηρόδρομοι ε, δεσμεύονται να σεβαστούν τα δικαιώματα ε, των επιβατών ε, και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επαρκή προστασία. Είναι σημαντικά τα δικαιώματα των επιβατών για μας. Θέλουμε λοιπόν μια λύση που να εγγυάται τα δικαιώματα αυτά και να επιλύει ενδεχόμενα προβλήματα. Γι' αυτό συμφωνούμε με κάποιε τροποποίησει, ε, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητε, Για παράδειγμα, όσον αφορά ε, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Και είμαστε βέβαιοι ότι ο μελλοντικό κανονισμό θα αποτελέσει πολύ καλή βάση για τα δικαιώματα των επιβατών. Πιστεύουμε όμως ότι χρειάζεται ακόμα να γίνουν κάποιες αλλαγές στο σχέδιο κειμένου που αντικατοπτρίζουν και τις αλλαγές που έχουν γίνει στον τομέα των σιδηροδρόμων. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λοιπόν τις πιο σημαντικές μας παρατηρήσεις. Άρθρο 2, κατά τη γνώμη μας, η διαγραφή των παρεκκλήσεων που προβλέπονται δεν θα είναι θετική, θα επηρεάσει πολύ τα ε, σχέδια ε, επενδύσεών μας και τον εξυγχρονισμό του τροχαίου υλικού. Σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε μεγάλο τμήμα του τροχαίου υλικού μας ε, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερο τροχαίο υλικό σε χρήση. οι νέες δημόσιες συμβάσεις για την αγορά και τον εξυγχρονισμό τροχαίου υλικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό είμαστε υπέρ της διατήρησης κάποιων παρεκκλήσεων. Δεύτερον, όσον αφορά το άρθρο 10, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τα ενιαία εισιτήρια, τα through tickets. Οι σιδηρόδρομοι ήδη συνεργάζονται μεταξύ τους σε κάποιες συμβάσεις και μπορούν έτσι να λαμβάνουν υπόψη τους καθυστερήσεις κλπ. Ε, η τροποποίηση, η πρόταση του άρθρου 6 μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όσον αφορά την υποχρέωση παροχής ε, πληροφοριών στους ε, επιβάτες ε, ή την ευθύνη. Και αυτό πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να κυριαρχήσει η αγορά. Επίσης, στο άρθρο 17 πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμη η ρήτρα αυτή. Πιστεύουμε όμως ότι είναι πολύ περιορισμένος ο ορισμός. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους ε, ενιαίους κανόνες ε, CIV, της Διεθνούς ε, Σύμβασης Μεταφοράς Επιβατών. Αυτά όσον αφορά την ανωτεραβία. διότι έτσι θα υπάρχει ασφάλεια δικαίου, θα αποφύγουμε τον κίνδυνο διαφορετικών ερμηνεών και θα έχουμε σταθερέ προποθέσει για τον ανταγωνισμό. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία και όσον αφορά ε, τον σχεδιασμό αντιμετώπιση ε, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ε, στο άρθρο 18.6. Η εκπόνηση τέτοιων αναλυτικών σχεδίων για τους σταθμούς θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας ε, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ε, κάποιες γενικές ε, διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, άρθρο 22, αρρωγή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παρέχεται συνδρομή 24 ώρες ε, την ημέρα, κάτι που δεν θα είναι δυνατό να γίνει σε όλους τους σταθμούς και αυτό θα οδηγήσει σε δυσανάλογο και αδικαιολόγητο κόστος. Άρθρο 26. Κατάρτιση του προσωπικού. Ήδη παρέχουμε τέτοια κατάρτιση. Δεν είναι όμως απαραίτητο αυτό να παρέχεται σε όλο το προσωπικό, μόνο στα άτομα που θα έχουν επαφή σε άτομα με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα. Συνοψίζοντα, ε, ήδη ο σιδηροδρομικό τομέα έχει επενδύσει σημαντικά για να ανταποκριθεί στι απαιτήσει ε, του ισχύοντο κανονισμού 1371 2007 που τέθηκε σε ισχύ το 2009. Αυτή τη στιγμή επενδύουμε στον εξυγχρονισμό του τροχαίου υλικού και των ε, σταθμών. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και των προϊόντων που ε, παρέχουμε στους επιβάτες, ε, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται λοιπόν η ισορροπημένη προσέγγιση ε, θα πρέπει να σεβαστούμε απολύτω τα δικαιώματα των επιβατών, από την άλλη θα πρέπει να επιβάλλουμε ρεαλιστικέ απαιτήσει στον τομέα. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, για, τους, για τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις εργασίες τους ε, σχετικά με την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών χωρίς να, διακινδυνεύεται, χωρίς να διακυβεύεται ο ανταγωνισμός του τομέα. Θέλουμε λοιπόν ε, συστήματα μεταφορών ε, φιλικά προς το περιβάλλον και χρειαζόμαστε επιπλέον οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του ε, πολιωτούς δημοσιονομικού πλαισίου και, του, και της, μετά το 2020 και της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κιντόρ έχει το λόγο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ε, εθνικών μεταφορών. Σας καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο για έξι λεπτά. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Επίσης θα ήθελα να, ε, να ζητήσω συγγνώμη από τον πρόεδρό μας, από τον Μπρούνο Γκαζό, ο οποίος θα έπρεπε να είναι στη θέση μου, αλλά πρέπει να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό για τον καινούριο νόμο για τους ε, σιδηροδρόμους. Η ΦΝΟΤ έχει 160 οργανώσεις και 80.000 μέλη. Ε, προβλέπει την ε, προστασία των καταναλωτών και των επιβατών. Για την ΦΝΟΤ, ο πρώτος ε, κανονισμός αποτελούσε την ε, βάση για να λαμβάνουμε υπόψη τις αποζημιώσεις για τους επιβάτες. Το κείμενο αυτό ορίζει τις ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές, ιδιαίτερα τις κύριες συνδέσεις, και τις, αλλά οι περιφερειακές δεν λαμβάνονται υπόψη. Όμως παρέμεινε νεκρό γράμμα, διότι μόνο 23 από τα 28 κράτη-μέλη ε, εφάρμοσαν αυτό το κανονισμό το 1371. Γι' αυτό δυστυχώς τα κράτη και οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να βρούμε ε, ε, μία κοινή βάση έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός και εναρμόνιση ως προς τις σιδηροδρομικές εναέριες και οδικές μεταφορές. Το δεύτερο είναι ότι για τη ΦΝΟΤ θα πρέπει να υπάρχει ρυθμισμένος ανταγωνισμός, ρυθμιζόμενος ανταγωνισμός, όπως ορίζει το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, για να έχουμε καλύτερες παροχές και μεγαλύτερο δέλεαρ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Όπως ε, ορίζει το τέταρτο πακέτο. Ως προς το σχέδιο αναθεώρησης, το οποίο υποβλήθηκε αυτές τις ημέρες, ε, έχουμε ορισμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θα παραμείνω στις γενικές μόνο κατευθυντήριες γραμμές και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις περιφερειακές και τοπικές μεταφορές, καθώς και τις δημόσιες συμβατικές μεταφορές, γιατί δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη το 80% των επιβατών μας. Γιατί από τους 10 χρήστες οι 9 χρησιμοποιούν τις ε, περιφερειακές σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λοιπόν αυτούς τους ε, καθημερινούς χρήστες που μεταβαίνουν στην εργασία τους, στο πανεπιστήμιό τους, που είναι συνδρομητές και που δυστυχώς πρέπει να υποστούν ε, τις καθυστερήσεις ή τις ακυρώσεις που έχουν επίπτωση στην επαγγελματική τους εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμός. Ελπίζουμε λοιπόν να τα καταφέρει αυτός ο κανονισμός. Αναγνωρίζουμε και ένα άλλο σημαντικό σημείο σε αυτή την αναθεώρηση που αφορά το ενιαίο εισιτήριο που θα πρέπει να ισχύει παντού. Θεωρούμε ότι όλοι οι επιβάτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το μέσον και μέσα στα πλαίσια ενός ε, μονοπωλίου θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε υπόψη το ενιαίο εισιτήριο με τον τελικό προορισμό. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την εγγύηση, την ε, τελική εγγύηση του επιβάτη και να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων και τον δελεστικό τους χαρακτήρα για να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ε, των επιβατών για να μπορέσουν ε, να εργαστούν και να μεταβούν στην εργασία τους όπως πρέπει δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αυτοί οι επιβάτες έχουν καθυστέρηση μία με δύο φορές την εβδομάδα. Και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ε, καθημερινές μεταβάσεις των επιβατών. Αυτό σημαίνει ουσιαστική διαφάνεια σε επίπεδο ωραρίων και ποιότητας των υπηρεσιών. Χρειάζεται λοιπόν ακρίβεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και το ενιαίο εισιτήριο με διαφάνεια. Άρα φτάνουμε στο τρίτο θετικό σημείο της προσβασιμότητας στους σιδηροδρόμους σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, διότι ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζει θέματα κινητικότητας και θα πρέπει να υπάρχουν οι υποδομές στους σταθμούς για να μπορέσουν να κινηθούν οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσχέρειες. Τώρα, για τις μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές είμαστε απόλυτα σαφείς. Ιδιαίτερα για τις ε, ε, σιδηροδρομικές αυτές γραμμές υψηλής ταχύτητας δεν θα πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση πάνω από μία ώρα τη στιγμή που το όλο ταξίδι διαρκεί δύο ώρες. Υπάρχουν πολλά intercity και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Άρα θα πρέπει να μειωθούν οι καθυστερήσεις κάτω από 30 λεπτά. Ως προς την ανωτέρα βία, δεν θέλουμε να σταθούμε πολύ επ' αυτού θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες ανωτέρας βίας κατά τις μεταβάσεις και την χρήση των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών. Χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση για όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει είναι υπεύθυνε σε περίπτωση ανωτέρας βίας για να υπάρξουν ε, λύσεις ε, αντικατάστασης και για να βοηθηθούν οι επιβάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μεγάλες ε, οργανώσεις και ενώσεις που προωθούν τα συμφέροντα του καταναλωτή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις οργανώσεις αυτές στα πλαίσια της χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να δούμε ε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό τον ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ε, η κυρία Αντάντ έχει το λόγο. Είσαστε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που ασχολείται με θέματα κινητικότητας και αναπηριών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε την ε, τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της, του κανονισμού. Καλώ ορίζουμε την αναθεώρηση του κανονισμού από το Φόρουμ Αναπηρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι εκπληρώνει τι υποχρεώσει τη σε ό,τι αφορά τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία που στο άρθρο 9 απαιτεί σαφέστατα προσβασιμότητα στις μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία. Άρα ο τομέας αστυνομικό θεωρούμε ότι έχει ήδη κάνει πολλά για να βελτιώσει την προσβασιμότητα αλλά δυστυχώς για τα άτομα όπως εγώ ανεξάρτητη μετακίνηση ε, χωρίς πρώτερο προγραμματισμό δεν είναι ακόμα κάτι το δυνατόν. Και μέχρι να πετύχουμε λοιπόν το στόχο αυτό, εμείς εξαρτώμαστε ακόμα στα... σε βοήθεια, από βοήθεια για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας σε, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 1371 και σε, ότα, σε όσα έχει πετύχει τα τελευταία 10 χρόνια. Η πρόταση αναθερήση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πληρώνει κάποια σημαντικά κενά τα οποία παλιά δεν προβλεπόντουσαν στον αρχικό κανονισμό. Για παράδειγμα, είμαστε ε, ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι η προαστιακή και οι τοπικοί σιδηρόδρομοι έχουν καλύτερες προβλέψεις ε, πλέον και επίσης ε, πιστεύουμε και το τονίζουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση πρόβλεψη για αρρωγή σε άτομα αναπηρία και ιδιαίτερη εκπαίδευση και τα μέλη και οι στόχοι μάλλον των εθνικών σωμάτων εφαρμογής ε, είναι πλέον καλύτερα ορισμένα. Ωστόσο, ένα σημείο στο οποίο έχουν κάνει μεγάλη εκστρατεία τα άτομα με αναπηρία και δεν έχει ακόμα, ακόμα αντιμετωπιστεί είναι η... ο κανόνας πρώτης ειδοποίησης 14 ώρες που εξακολουθεί να παραμένει στην αναθεώρηση του κανονισμού δεν συνάδει αυτό με τη σύμβαση του ΟΗΕ και είναι εντελώ παροχημένο. Για παράδειγμα, αν το αφεντικό μου μου ζητήσει να πάω στο Παρίσι αύριο, είμαι υποχρεωμένη να αρνηθώ γιατί δεν έχω α, ε, κάνει κράτηση για βοήθεια. Ακόμα και αν βγω το βράδυ, για παράδειγμα, για να το δεν μπορώ να μείνω λίγο παραπάνω, γιατί αν μείνω παραπάνω δεν ε, μπορεί να έχω το τρένο για το οποίο έχω κάνει κράτηση, γιατί δάλλως δεν ε, θα με βοηθήσει κανένα να μπω στο τρένο για να γυρίσω στο σπίτι μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει προτεραιτητοποίηση, υποχρέωση προτεραιοποίηση. Στην Ολλανδία α, το διάστημα έχει μειωθεί σε μία ώρα για την προτεραιοποίηση και στην Δανία αυτή η προτεραιοποίηση πρόσφατα μειώθηκε στις 12 ώρες και ακόμα και εδώ στο Βέλγιο έχει μειωθεί στις 3 ώρες σε πιο πολλούς από 25 συνδρομικούς σταθμούς. Άρα το Ευρωπαϊκό Φόρμα Αναπηρίας ζητάει μια σαφή πολιτική προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ταξιδεύουν όπως όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες. Πέρα από αυτή τη βασική αξίωση, το μου θα ήθελε μια πιο λεπτομερή περιγραφή της εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού ε, ιδανικά θα θέλαμε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά την κατάρτιση αυτή για να υπάρχει πραγματικά καλό επίπεδο α, και καλή ποιότητα. Και τέλος θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται με τις συγκεκριμένες ε, αρμοδιότητες των σωμάτων εφαρμογής που δεν εξετάζουν μεμονωμένες καταγγελίες και δεν εναρμονίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα συνοψίζοντας το EDF υποστηρίζει το μεγαλύτερο τμήμα της πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Με χαρά την επιστώνουμε ότι υπάρχουν βελτιώσεις για τα άτομα με αναπηρία, αλλά πραγματικά θέλουμε να καταργηθεί αυτή η υποχρέωση πρώτη ειδοποίηση 48 ώρων και να βελτιωθεί η κατάρτιση του προσωπικού και να ενισχυθούν και οι αρμοδιότητες των εθνικών σωματών και των αστυνικών υπηρεσιών. Όσοι δεν ενδιαφέρονται πιο πολύ να λάβουν πιο πολλές πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρίες, την επόμενη εβδομάδα, 28 Φεβρουαρίου στις 1 ε, το μεσημέρι, το... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανωθεί μια σχετική εκδήλωση στην οποία και θα συμμετάσχει και το δικό μας φόρουμ, το EDF. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις διευκρινήσεις σας και να συνεχίσουμε με τον κύριο Σμιόλτερς μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Επιβατών. Έχετε το λόγο για έξι λεπτάκια και εσείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρε, την κυρία Ντελή, τον ε, εισηγητή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κοινό που μας ακούει. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βλέπετε εδώ τον χάρτη του EPF από τον, φέτος τον Φεβρουάριο. Έχουμε 38 οργανώ, οργανισμούς μέλη σε 21 χώρες, αυτές που φαίνονται με μπλε στον χάρτη. Ιδρυθήκαμε το 2002 και είμαστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εθνικών και Περιφερειακών Οργανώσεων Επιβατών. Σε κάποιες χώρες, ε, ανάλογα με τις περιφέρειες και όλα, ε, μπορεί να έχουμε πάνω από μία ε, οργάνωση χρηματοδοτούμαστε από τα μέλη μας, ε, από τις οργανώσεις μέλη μας, αυτό είναι το μόνο μας ε, έσοδο αυτή τη στιγμή και εκπροσωπούμε τις απόψεις επιβατών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολούμαστε με όλα τα είδη μαζικών μεταφορών, όπως είναι οι τοπικές μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι, τα λεωφορεία, τα αεροπλάνα και τις θαλάσσιες μεταφορές όσον αφορά τις πληροφορίες και την ευθύνη. Πιστεύουμε ότι τα εισιτήρια που πολλούνται πρέπει να έχουν εγγύηση μέχρι τον τελικό προορισμό, δηλαδή ε, εγγύηση ενιαίου εισιτηρίου. Πιστεύουμε ότι ε, πρέπει να επιβληθούν περισσότερες ε, υποχρεώσεις στους πολιτές εισιτηρίων, στους φορείς τους διαχειριστές των υποδομών και τους υπεύθυνους ε, σταθμών. Και ε, θα πρέπει να ισχύουν οι απλοί κανόνες του ενοχικού δικαίου. Ε, ο οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται το προϊόν που έχει πωλήσει και θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα στους σταθμούς της τους σταθμούς, τα τρένα και τις αποβάθρες, ε, διότι στο Βέλγιο μπορεί να είναι προσβάσιμος ο σταθμός, ε, όχι όμως ε, η αποβάθρα. Χρειάζεται λοιπόν πιο εύκολη πρόσβαση για όλους, διότι και η Ευρώπη γυράσκει και οι γέροι έχουν συχνά περιορισμένη κινητικότητα. Εάν γίνει αυτό, αυτό θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των επιβατών. Εάν δεν μπορεί να παρασχεθεί αυτό, χρειαζόμαστε τουλάχιστον ε, μια προειδοποίηση το αργότερο 24 ώρες πριν. Ε, θέλουμε σε συνθήκες ανταγωνισμού για όλα τα είδη μεταφορών. Υπάρχει παρέκκληση για περιφερειακούς και προαστιακούς ε, σιδηροδρόμους ε, και η έκθεση της UITP έδειξε ότι το 90% των ταξιδιών των, ε, επιβατών και το 50% όσον αφορά την απόσταση σε χιλιόμετρα γίνονται σε τοπικά συστήματα και νομίζω ότι σημαντικό είναι ότι κάποιοι φορείς ε, ήδη σήμερα συμπεριφέρονται στον επιβάτη σαν να είναι βασιλιάς. Ε, ε, πριν τέσσερα χρόνια απένιμα βραβείο στην επιχείρηση North Αφεκίας Φεαποντ και η επιχείρηση αυτή, εάν υπάρξει πεντάλεπτη καθυστέρηση στο τελικό προορισμό, επιστρέφουν τα χρήματα. Υπάρχει εγγύηση για ε, τις συνδέσεις ακόμη και το βράδυ. Ε, και υπάρχει εγγύηση για τις υπηρεσίες, για την παροχή πληροφοριών, για ε, την φιλικότητα προς τον επιβάτη. και ξέρω ότι αυτό θα ασκήσει πίεση στους ε, συνδρομικούς φορείς. Σήμερα όμως με την ψηφιοποίηση μπορεί να υπάρξει απόλυτος έλεγχος της λειτουργίας. Και η επιχείρηση που σας έδωσα όχι μόνο ε, επιχείρηση, αλλά αποτελεί και πολύ καλό παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την ανωτέρα βία, ο ισχύων κανονισμός κατόπιν της απόφασης του, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γενικά είναι ε, φιλικός προς τον πελάτη. Γενικά λαμβάνει το 50, αποζημίωση του ε, 50% του, της τιμής του εισιτηρίου το πολύ. Ε, οι συνδρομικοί φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ε, και να παρέχουν ε, βοήθεια στους επιβάτες που δεν έχουν φτάσει στον τελικό προορισμό τους. Και γενικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση τώρα να παρέχουν πληροφορίες. Και φτάνω τώρα στην τελευταία μου διαφάνεια πριν την σύνοψη. Βλέπετε εδώ μια μικρή εικόνα του Δαβίδ και του Γολιάθ που δείχνει τον επιβάτη σε σχέση με τη συνδρομική επιχείρηση. Σήμερα οι ε, οργανώσεις επιβατών ε, δεν έχουν ε, αρκετή ισχύ και όχι επαρκές προσωπικό και συχνά είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση οι επιβάτες στους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Χρειάζεται λοιπόν υποχρεωτική εναλλακτική επίλυση διαφορών για τους επιβάτες. Ε, η Οδηγία 2013-11 για την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν είναι επαρκώς γνωστή στους πελάτες. Γενικά θα πρέπει να παρακολουθείτε η ικανοποίηση των επιβατών. Σήμερα ήδη το βλέπουμε αυτό στο Travel Watch Southwest, το London Travel Watch κλπ. Ε, το EPF θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει αυτό το ρόλο μέσω των τοπικών μας οργανώσεων. Και φτάνω στην ε, σύνοψη της ε, της ομιλίας μου να παραμείνει το θέμα της ανωτέρας βίας όσο έχει σήμερα, να συμπεριληφθούν οι περιφερειακές και προαστιακές ε, σιδηροδρομικές γραμμές, ε, να υπάρχει εγγύηση ενιαίου εισιτηρίου, να βελτιωθεί η προσβασιμότητα όταν δεν υπάρχει να δίδεται προειδοποίηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν και να παρακολουθείτε η ικανοποίηση των επιβατών. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Ρέφεν ο οποίος είναι υπεύθυνος στα πλαίσια του, στο ρυθμιστικό πλαίσιο των σιδηροδρόμων στη Δανία. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Υποστηρίζουμε την πρόταση, απλώς έχουμε ορισμένες ε, επιπλέον προτάσεις για βελτιώσεις. Καταρχήν, οι ορισμοί που έχετε. Στην, στο άρθρο 10, παράγραφος 5, μιλάτε για ticketing machine, αλλά δεν έχουμε κανέναν ορισμό στην ε, πρόταση. Τι είναι αυτή, αυτό το μηχάνημα πώληση εισιτηρίων. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν ορισμό για το ticketing machine και επίσης θεωρήσαμε ότι αυτός ο ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει την ε, κάρτα ταξιδίου. Στη Δανία έχουμε ένα τέτοιο σύστημα έκδοσης καρτών που λειτουργεί πάρα πολύ καλά στη Δανία όπως και σε άλλες. Κύριε Σμέλντερς, μπορείτε να... Α, εντάξει, ωραία, κλείσατε το μικρόφωνο σας, γιατί γίνονται παρεμβολές. Προτείνω λοιπόν να εισαγάγουμε έναν ορισμό για το τι σημαίνει ticketing machine και σε αυτό τον ορισμό να λάβουμε υπόψη και τις ε, κάρτες ταξιδίου. Έτσι, να μην υπάρχει ε, φόρτος επιπρόσθετος φόρτος για τους σιδηροδρόμους, γιατί οι παραδοσιακές, τα παραδοσιακά μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων είναι πιο, ε, δίνουν πιο ακριβά εισιτήρια από τις κάρτες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Κατά την άποψή μας, αν ε, δείτε ποιες είναι αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων. Είναι πολύ χαμηλές οι αποζημιώσεις αυτές. Εάν υπάρχει καθυστέρηση μίας και δύο ώρων, έχετε 25% αποζημιωση Αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τόσο χαμηλό που πολλές φορές δεν γίνεται καν αίτηση αποζημίωσης από τους ενδιαφερόμενους. Και εδώ βλέπετε τις ποσοστιαίες αναλογίες που ισχύουν στην επικράτεια της Δανίας. Άρα προτείνουμε να αυξηθούν αυτά τα ποσοστά αποζημίωσης. Έτσι θα, θα μειωθεί η έλλειψη ικανοποίησης επιβατών σε, για λόγους καθυστέρησης και θα αποφευχθούν και οι καθυστερήσεις. Προτείνουμε λοιπόν να αυξηθούν οι ποσοστιαίες ε, αναλογίες αποζημιώσεων. Στη συνέχεια, στο άρθρο 18, παράγραφο 2α, υπάρχει αυτή η υποχρέωση για τους σιδηροδρόμους, ε, για ε, καθυστερήσεις άνω των 60 λεπτών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρέπει να ε, υπάρχει παροχή τροφίμων και ποτών για τους επιβάτες. Και αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον προμηθευτή. Εμείς προτείνουμε να απαλείψουμε το κόκκινο, δηλαδή την φράση αυτή την υπογραμμισμένη με κόκκινα, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει υποχρέωση έτσι κι αλλιώς ε, παροχής ε, τροφής. Και θα πρέπει να σκεφτείτε έμπρακτα την κατάσταση. Κάπου ε, έχει σταματήσει το τρένο και όλοι προσπαθούν να το θέσουν εν κινήσει. Δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η υποχρέωση της επιχείρησης ε, να παρέχει σάντουιτς και ποτά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν τη στιγμή που έχει σταματήσει το τρένο. Πρέπει να στείλουν, να στείλουν τι, κάποιον να πάει να βρει αυτά τα τρόφιμα και τα ποτά. Θα πρέπει να παρασχεθούν δωρεάν στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από τη μία ώρα, τότε ο επιβάτης μπορεί να δώσει μία απόδειξη για τις δαπάνες και να αποζημιωθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ώστε η επιχείρηση να παρέχει σάντουιτς και ποτά. Δεν έχει νόημα αυτή η πρόταση. Προτείνουμε δηλαδή το κόκκινο να απαλληφθεί. Επίσης, ε, και πολύ το προανέφεραν και συμφωνώ, υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες ε, είναι υπερβολικές δηλαδή να υπάρχει παροχή βοηθείας στις αποβάθρες ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή στους σταθμούς. Πρόκειται για τις υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων 22 και 23. Νομίζω ότι είναι υπερβολικές αυτές οι απαιτήσεις. Και δεν έχει νόημα για παντού, γιατί στη Δανία η είσοδη προς τα τρένα, στα τρένα ε, είναι εξοπλισμένες για αυτούς δηλαδή που θέλουν να μπουν με αναπηρικά μαξίδια και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η απέτηση. Θα ήθελα να φτάσετε στα συμπεράσματά σας. Ναι, το τελικό άρθρο είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση προς τους επιβάτες ως προς τα δικαιώματά τους. Και εδώ έχουμε ορισμένες ε, προτάσεις τροποποίησεων. Θα πρέπει να ορίσουμε αυτές τις υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση. Γιατί αν δεν αναφέρονται ρητά, δεν υπάρχουν. Νομίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κενά. Θα πρέπει να αναφερθούμε και στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και αυτό στους επίσημους ιστοτόπους των σιδηροδρόμων. Τέλος, στη Δανία οι πληροφορίες παρέχονται από μεγάφωνα σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα θέλαμε αυτό να προστεθεί στις υποχρεώσεις. Στο παράθεμα επίσης 2 Υπάρχει ένα παράρτημα με ελάχιστε πληροφορίες από τις επιχειρήσεις και τα σημεία, για τα σημεία πώλησης ε, εισιτηρίων. Το άρθρο 30 θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε αυτό το δεύτερο παράρτημα. Θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας, ε, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο κύριο Μάρκ Σμιθ. Πού είστε, πού κάθεστε, ωραία. Ήρθατε με το γιο σας. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι ο γιος σας. Α, εκεί, εκεί. Είδε να δει, ήρθε να δει πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλει, ας έρθει να καθίσει δίπλα μου. Έλα να καθίσεις δίπλα μου. Από εδώ θα βλέπεις καλύτερα. Μη φοβάσαι. Ίσως είσαι ένας μελλοντικός ευρωβουλευτής. Il est très impressionné. Bienvenue. Tu me donnes ça? Ah, think he is. Ναι, φυσικά, φυσικά να τον χειροκροτήσουμε. Βάλε και τα ακουστικά σου. Number two. Okay. Okay, great. Bon, alors, nous avons donc... Έχουμε έναν ε, α, νέο συνάδελφο μεταξύ μας και ας ακούσουμε τον κύριο Σμιθ. Είσαστε blogger στο blog SEAT61. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Για 6 λεπτά. Έχετε το λόγο. Well, good morning Καλημέρα σε όλους σας και σας ευχαριστώ που καλέσατε εμένα και το γιο μου ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι ως blogger και έχω ε, μια ιστοσελίδα ε, που βοηθάει τους ανθρώπους να ταξιδεύουν στην Ευρώπη με το τρένο. Κάθε μέρα ασχολούμαι με τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών και έχω και την τύχη να ακούσω και τις απόψεις των νομοθετών επί του θέματος γιατί παλαιότερα εργαζόμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και η δική μου η ομάδα ήταν εκείνη που εξέδωσε ρυθμίσει ε, σχετικά με το συνδρομικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουμε 20 διαφορετικούς φορείς. Ε, και παλαιότερα εργαζόμενος μάνατζερ, manager. Γνωρίζω λοιπόν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ε, να υπάρχουν όλες αυτές οι εξελίξεις για του σιδηροδρόμους. Κατά τη δική μου άποψη το μεγαλύτερο θέμα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιβάτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους είναι αυτό που θεωρώ ως ο κίνδυνος 500. Ε, θα εξηγήσω ένα, με ένα παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι μια οικογένεια ζει στο Όστεμπουργκ και θέλει να πάει στο Παρίσι για Σαββατοκύριακο. Ο πιο σύντομο δρόμο είναι Deutsche Bahn στην κολονία Ταλή ε, στο Παρίσι. Ε, Deutsche πάνω ε, από την κολονία ε, έχει ένα 19,90 ευρώ, κατόπιν 35 ευρώ στο τελή, σε πολλά χρήματα, 3 ε, ώρες 30 λεπτά η ε, διαδρομή. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι αδύνατον στο σημερινό, σημερινή κατάσταση να αγοράσει κανείς ένα δωρεάν εισιτήριο. Παλαιότερα ήταν δυνατόν, σήμερα δεν είναι πια. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν αγοράσει, αγοράσει κανείς ε, αυτό το εισιτήριο σε μια ιστοσελίδα, παρότι μια να είναι μία συναλλαγή, αποκτά κανείς δύο εισιτήρια. Ε, δύο εισιτήρια λοιπόν που σημαίνει και δύο συμβόλαια. Ε, βεβαίως όλα είναι καταπληκτικά αν πάνε στην ώρα τους, ε, αλλά αν τελικά αργήσει το, η Deutsche Bank και χάσει κανείς το τελίστη θα γίνει. Αυτό το ξερτισμένη την έχει πατήσει κανείς, ας το πούμε απλά. Και το λέω αυτό διότι οι εταιρείε αυτές ε, έχουν ε, πολύ καλή φήμη. Ε, πολλές εταιρείε λένε είμαστε ξεχωριστή εταιρεία, λέει Ταλής, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την Deutsche Bahn, ε, τώρα το εισιτήριό σας των 35 ευρώ ε, δεν έχει καμία αξία και αν θέλετε να πάτε στο επόμενο δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, 122 ευρώ είναι το επόμενο εισιτήριο αν θέλετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας για το Παρίσι. Ως εκ τούτου η επιλογή που υπάρχει είτε να δώσει κανείς 500 ευρώ και να συνεχίσει το ταξίδι ή να πάνε πίσω σπίτι τους ε, και ε, να ε, γλιτώσουν ε, χρήματα από το τρένο, αλλά θα πληρώσουν αυτά που θα πλήρωναν στο ξενοδοχείο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σωστά. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η ασφάλεια των τρένων δεν καλύπτει αυτήν την περίπτωση, γιατί και αυτή είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Ως εκ τούτου, για άλλη μια φορά, πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά στους ε, επιβάτες. Βεβαίως, αν το τρένο της Deutsche Bahn αργούσε μία ώρα, ε, θα έπαιρνε κανείς πίσω 20 ευρώ. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε εδώ να μιλάμε για τον κίνδυνο των 480 ευρώ, αντί για 500 ευρώ. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένος ε, ότι το κοτήφε CV δεν είναι πια καλό, δεν μας ταιριάζει, ε, και λέει ότι αν χάσει κανείς το επόμενο τρένο ε, τότε ε, υποτίθεται δεν θα πληρώσει για το επόμενο τρένο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όμως το CIV παλαιότερα όταν ήταν μόνοι τους αυτοί βγάζουν δύο εισιτήρια. Εγώ παλαιότερα έπρεπε ας πούμε για το Λονδίνο στο, στην Κωνσταντινούπολη να έχω τρία εισιτήρια και Αυτά όμως έχουν παρέλθει πλέον. Η προστασία δεν ισχύει όταν έχουμε δύο εισιτήρια ε, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όμως χρειάζεται κανείς προστασία. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν τα δύο εισιτήρια υπάγονται στην CIV, η προστασία που υποτίθεται ότι προσφέρεται, η προστασία αυτή κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί. Αν πάμε πίσω σε μονολυθική βασικούς εθνικούς ε, ε, φορείς το πρόβλημα εξαφανίζεται. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Και αν θέλουμε μια δυναμική σιδηροδρομική αγορά, το πρόβλημα θα γίνει μεγαλύτερο με περισσότερους φορείς, περισσότερα ξεχωριστά εισιτήρια ε, και περισσότερους που θα χρησιμοποιούν συνδυασμό εισιτηρίων για να προγραμματίσουν το ταξίδι τους. Και πιστεύω βέβαια ότι υπάρχει μια αρκετά απλή λύση. Δηλαδή να αναθεωρήσουμε το CIV για τον 21ο αιώνα ε, την προστασία να την προσφέρουμε σε όλους τους επιβάτες ανεξάρτητα από το αν οι επιβάτες έχουν από ένα έως και τρία εισιτήρια. Το 2017 οι διάφοροι εθνικοί φορείς ε, συνεργάστηκαν και υπέγραψαν μια εθελοντική συμφωνία για τη συνέχιση του ταξιδιού που κάνει ακριβώς αυτό. Έχω δει τη διατύπωση, είναι απλή, δεν είναι γραφειοκρατική, δεν νομίζω ότι κοστίζει τίποτα. Ε, απλά ε, βγάζει κανείς επόμενο εισιτήριο για την επόμενη διαδρομή επειδή ένα τρένο έχει καθυστορήσει και το γεγονός ότι έχει υπογραφεί μια εμπορική συμφωνία καταδεικνύει ότι τελικά ε, πράγματι αυτό είναι και προς το συμφέρον της εταιρείας μεταφορών. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την βελτίωση και την επέκταση της Ευρώπης ε, να έχουμε ένα δίκτυο, να μην έχουμε αποκομμένους ε, φορείς. Ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και να προστατεύουμε τους επιβάτες να κάνουν και τρία εισιτήρια ανεξάρτητα και τρία ταξίδια ανεξάρτητα το πώς έχουν εκδοθεί τα εισιτήρια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σμιθ. Ο κύριος Λόχμαν είναι ο, ο τελευταίος ε, παρεμβαίνων. Είσαστε υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Υποδομών Σιδηροδρόμων, της CER. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας ε, για ε, τα δικαιώματα των επιβατών ε, σε κάποια θέματα. Εδώ βλέπετε ποια είναι τα μέλη μας. Είναι οι εκπρόσωποι των συνδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών των υποδομών. Εκπροσωπούμε λοιπόν το 93% του τομέα αυτού, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε για τις προσδοκίες ε, των επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Οι επιβάτες ε, είναι οι πελάτες μας άλλωστε. Τι σημαίνουν για μας τα δικαιώματα των επιβατών. Μπορούμε να πάμε και πιο πίσω από το 2007 που είχαμε την πρώτη ρύθμιση των ε, δικαιωμάτων των επιβατών, διότι Είχαμε δικό μας χάρτη επιβατών που διαπραγματεύτηκαν τα μέλη της Ένωσής μας που είχαν ε, την διάθεση να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους επιβάτες. Και μάλιστα ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών ε, ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια αυτό που έκαναν οι επιχειρήσεις μας σε θελούσια βάση. Συνεχίζουμε να έχουμε επαφές ε, με ε, ευρωπαϊκές ενώσεις επιβατών και καταναλωτών και έχουμε ε, σε τακτική βάση συνάντηση με αυτούς ώστε να έχουμε εικόνα των προσδοκιών των επιβατών και των δυνατοτήτων βελτίωσης των υπηρεσιών. Ε, άλλωστε είναι προ συμφέρον ε, των ε, επιχειρήσεων να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και στην εικόνα αυτή βλέπετε διάφορα στοιχεία που πιστεύουμε ότι λειτουργούν αρκετά καλά συμπεριλαμβανομένων όπως είπα στην αρχή της συνεργασίας μας με τις ενώσεις επιβατών και με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Σίγουρα λοιπόν μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε το συμφερόν του επιβάτη. Τι περιμένουμε λοιπόν από την αναδιατύπωση του κανονισμού. Βελτίωση για τους πελάτες ε, χωρίς δυσανάλογα μέτρα για τις ε, επιχειρήσεις σιδηροδρόμων. Δηλαδή να έχουμε ε, ανταγωνιστικό περιβάλλον σε σχέση και με όλα τα είδη μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των επιβατών και της επιχειρήσεις μας. Αναφέρθηκε πολύ, πολλές φορές σήμερα το ενιαίο εισιτήριο, το through ticket και πολύ χάρηκα που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την αρχή ότι δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε νέες υποχρεώσεις αλλά να παρέχονται οι σωστές πληροφορίες. Ε, ποια ποιο είναι το συμβόλαιο, ποια είναι η σύμβαση που διέπει το ενιαίο εισιτήριο. Ιστορικά είχαμε διασυνοριακή συνεργασία, σήμερα έχουμε πιο ανταγωνιστικές αγορές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει στον τομέα των αερομεταφορών ή των ε, οδικών μεταφορών των λεωφορείων. Χρειάζεται λοιπόν συνεννόηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις ε, που συμμετέχουν στη μεταφορά. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε την αρχή του ενιαίου εισιτηρίου στα λεωφορεία και να μην το έχουμε ε, στα αεροπλάνα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε συνεργασία ανάμεσα στην Air France και την Ryanair. Θέλουμε λοιπόν ε, να εργαστούμε περισσότερο πάνω στο θέμα του ενιαίου εισιτηρίου, θα πρέπει όμως να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό για μας σήμερα και τι κάνουμε ήδη σήμερα. μετά από την εφαρμογή κανονισμού αλλά και πριν ε, είχαμε αναπτύξει ένα μοντέλο through service ενιαίου εισιτηρίου που δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν με ένα κλικ το εισιτήριο για όλη τη διαδρομή τους. Βλέπετε το παράδειγμα στην ε, οθόνη σας ε, μέσω της το τσεμπάν μπορεί να αγοράσει κανείς εισιτήριο από το Αμβούργο στην Ρώμη ή σε κάποιο μικρό χωριό της Αυστρίας. Χάρη λοιπόν στο μοντέλο αυτό που έχουμε εφαρμόσει σχετικά σύντομα, ε, έχουμε ε, κάτι το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τον κανονισμό. Κατόπιν ε, έχουμε το θέμα των επιβατών που δεν έχουν φτάσει στον τελικό τους προορισμό για τις υπηρεσίες υψηλή ταχύτητα υπάρχει υποχρέωση για την επιχείρηση να αναλάβει τους επιβάτες σε περίπτωση προηγούμενη καθυστέρησης, ακόμα και αν αυτή προκλήθηκε σε άλλη εταιρεία. Και επίσης υπάρχει υποχρέωση συνόχισης ε, του ταξιδιού ε, για κάθε είδος τρένου, αλλά όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω πριν, πρόκειται για συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων για τους πελάτες των επιχειρήσεων αυτών. Η συμφωνία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πιλωτική φάση. Θα πρέπει λοιπόν να την επεξεργαστούμε περισσότερο. Δεν πιστεύουμε όμως ότι αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί νομικά, διότι δεν ρυθμίζεται σε άλλους τομείς, όπως είναι οι οδικές μεταφορές, τα αεροφορία δηλαδή, ή, τα... ή οι αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανοίγουμε τη συζήτηση, αλλά πριν υπενθυμίζω πώς λειτουργεί η μέθοδος ping-pong. Είναι πολύ απλό. Στον πρώτο γύρο θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις και στο δεύτερο γύρο, σε όλα τα μέλη που θέλουν το λόγο, έχετε πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά να μας πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας. Γι' αυτό διαχειριστείτε καλά το χρόνο σας, γιατί δεν θα έχετε περισσότερο. Σας ε, κοιτάω κατά πρόσωπο, κύριε Μισουργέ, αλλά αυτό το κάνω γιατί είστε το πρώτος. Είστε έτοιμος. Έχετε το λόγο θα μας πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας και μετά θα υποβάλλετε την ερώτηση. Η κυρία Άντερσον. Θα έχουμε το λόγο πριν, γιατί είμαστε εισηγητές. Ο κύριος Λιμπεράτσκι πρέπει να φύγει, αλλά δεν έχει πέντε λεπτά. Γιατί εγώ τον αντικαθιστώ. Ναι, ο κύριος Λιμπεράτσκι μου είπε ότι φεύγει, αλλά αν τον, ε, έχετε, αν τον αντικαθιστάτε τότε θα έχετε φυσικά το λόγο για πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά για την κυρία Άντερσον. Ωραία, έχετε το λόγο. Καταρχήν, στην περίπτωση της ανωτέρας βίας θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συνδυροδρόμων κατά πόσο θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εξαίρεση. Εάν υπήρχε εξαίρεση, τότε θα δημιουργούσε μεγάλη νομική ανασφάλεια, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ αρνητικό για την επιχείρηση. Είναι αυτό ένα θέμα. Επίσης, το κύριο Λόχμαν θα ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο οι επιχειρήσεις σιδηραδρόμων μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Γιατί πολλοί επιδοτούνται εδώ και πολλά χρόνια από τους επιβάτες και τους φορολογούμενους. Γι' αυτό θα πρέπει να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων δεν θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω τον Πολωνό συνάδελφο από τους πολωνικούς σιδηροδρόμους κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση για θέματα αναπηριών. Θα μπορέσετε να, να υποβάλλετε όλες τις ε, ερωτήσεις, αλλά θα πρέπει να δώσετε και το λόγο να απαντήσουν οι πάνελιστ. Ως προς τις αναπηρίες, γιατί θα πρέπει να εκπαιδεύονται όλοι, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα πρέπει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα. Λυπάμαι που δεν σας άφησα πολύ χρόνο. Ωραία. Από ποιον αρχίζουμε. Μιλήσατε για την ε, ανωτέρα βία καταρχήν. Το συζητήσαμε στις αρχές του μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρούμε ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος σε σχέση με τις σημερινές προτάσεις. Δηλαδή, το καλύτερο θα ήταν να παραμείνουμε στο status quo. Ευχαριστώ. Πράγματι ε, πάντα μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα, αλλά εγώ θέλω να πω σχετικά με την ερώτηση αν υπήρχε καλή χρηματοδότηση, να πω ναι σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και ε, θα ήταν μια τεράστια διαφορά ε, αν κάναμε διαφοροποίηση ανάμεσα στους 14 και τους 13. Στους 13 σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι τραγική, άρα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί την παροχή υπηρεσιών. 64% είναι αποζημίωση. Εάν λοιπόν καταργήσουμε τις εξαιρέσεις και θεωρήσουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η παροχή των υπηρεσιών, πρέπει να εμπλακούν και οι αρμόδιες αρχές. Και μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει βελτίωση, χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Monsieur Olszewski, vous répondez Κύριε Ολσέσκι, θα απαντήσετε. E, Όταν πρόκειται για την εκπαίδευση του προσωπικού, Ε, υπάρχει, προβλέπεται κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα για αυτούς που ασχολούνται με την ασφάλεια του χώρου έχουν την ε, κατάλληλη κατάρτιση ε, υπάρχει και μία ειδική γραμμή βοήθειας όπου μπορείτε να καλέσετε για βοήθεια στο σταθμό ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Επίσης, ε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι λειτουργεί το σύστημα Anderson. Άλλη μία ερώτηση. Ο συνάδελφος από τη Δανία της ε, ρύθμισης σιδηροδρόμων δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι εθνικοί οργανισμοί εφαρμογής και ρύθμισης, ότι χρειάζεται δηλαδή επιπρόσθετη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Thank you. Ε, well... Σας ευχαριστώ πολύ το να αυξήσουμε τι αρμοδιότητε των ρυθμιστικών αρχών είναι καλή ιδέα, αλλά ειδικά στη Δανία δεν έχουμε το πρόβλημα αυτό, διότι η νομοθεσία μας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία. Δεν είναι λοιπόν πρόβλημα για μας, καταλαβαίνω όμω αυτό που λέτε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Ρενό Μεζολιέ, η Προς τον κύριο Κιντό, Κιντό ε, απευθύνω την πρώτη ερώτηση. Μιλάτε για το ενιαίο εισιτήριο. Κύριε Μιζολιέ, έχετε πέντε λεπτά. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε με αυτή την ταχύτητα για τους διερμηνείς. Ναι. Είναι επειδή δεν έχουμε χρόνο. Ναι, αλλά πρέπει να σέβεστε και τους εργαζόμενους. Κύριε Κιντόρ, ευχαριστούμε, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας ε, και εγώ τάσομαι υπέρ του ενιαίου εισιτηρίου και μιλάμε βεβαίως και για μέγιστη καθυστέρηση μισής ώρας, να περάσουμε από τη μία ώρα στη μισή ώρα. Υποστηρίξατε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις τοπικές σιδηροδρομικές γραμμές και τις περιφερειακές. Συμφωνώ. Τι θα πρέπει όμως να προσθέσουμε για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει ενίσχυση του ανταγωνισμού σε αυτό το επίπεδο, ναι ή όχι. Και όλα αυτά τα είπα σε 45 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ τον Ευρωβουλευτή. Βεβαίως ο ανταγωνισμός βοηθά ε, στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Καθίσταται σαφές ότι χρειάζεται βελτίωση παροχών υπηρεσιών που θα πρέπει να βασίζεται στο κόρπους των δικαιωμάτων των ε, επιβατών. Και φυσικά έχουμε και ολοένα και περισσότερους χρήστες που τίνουν προς το ναι. Ως προς τις τοπικές υπηρεσίες, κύριε Μιζολιέ, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση θα πρέπει να μιλάμε για τις ε, περιφερειακές ε, μεταφορές σε διάκριση με τις τοπικές. Γιατί αυτό που έχει σημασία ε, είναι να δούμε για, του, τα αμαία πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα όπως είναι αυτό του μετρό του Λονδίνου, του Παρισιού και του Βερολίνου. Και θα πρέπει να τονίσω ότι πολλοί από αυτούς είναι συνδρομητές. Δεν πληρώνουν ένα ή δύο ευρώ, α, καταβάλουν εκατοντάδες ίσως και, ίσως και χιλιάδες ευρώ ετησίως. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει προστασία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να τους ξεχάσει ο νομοθέτης. Ευχαριστώ κύριε Κιντόρ. Λόχμαν, κύριε Λόχμαν, μόνο τέσσερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό του 2007 χωρίς εξαιρέσεις. Πώς από το 2019 θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο κανονισμός. Γιατί υπάρχουν 2.024 εξαιρέσεις που προβλέπονται. Και τι θα γίνει στον ορίζοντα που θα μας οδηγήσει από το 19 μέχρι το 25 και μέχρι το 2030. Νομίζω ότι αυτή είναι ερώτηση περισσότερο προς τα κράτη-μέλη. Ε, αλλά δεν ε, υπερασπιζόμαστε καμία παρέκκληση και αναφερόμαστε σε αυτές μόνο σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση της υποδομής ή των ε, οχημάτων ε, δεν μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε σωστά τον κανονισμό. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Okay. Αλλά πρέπει να ισχύσει και να εφαρμοστεί από το 2019. Γι' αυτό ακριβώς και το ανέφερα στην ε, κυρία Χαντάντ. Θα ήθελα να πω τα εξής. Είπατε ότι πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες είναι αποτελεσματικές. Στην, ε, σε επίπεδο κομισιών υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης στους σταθμούς ιδιαίτερα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα αμαία και τους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα γενικότερα. Αλλά πώς θεωρείτε ότι εξελίσσεται αυτό το επίπεδο. Ναι, μιλάμε 15% του πληθυσμού. Εμείς μιλάμε για τα δικαιώματα 80 ε, εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας. Έχω δικαίωμα για άλλη μια ερώτηση. Κύριε Σμιθ, κατά την πείρα σας στις περιπτώσεις καθυστέρησης ή ε, αναβολής, πώς τηρούν τα δικαιώματά τους και τι ανταπόκριση υπάρχει, ιδιαίτερα σε περίπτωση ακύρωσης. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ενημερώνει κανείς ε, τους επιβάτες για τα δικαιώματά του σε περίπτωση καθυστέρηση ήδη στην αρχή του ταξιδιού, διότι εάν κάποιος ε, όταν πουλάει ένα προϊόν ε, του λέει τι μπορεί να πάει στραβά, δεν είναι πολύ καλός πολιτή. Το θέμα είναι ότι μεγάλο τμήμα του προσωπικού δεν γνωρίζει αρκετά καλά τα δικαιώματα των ε, επιβατών και χαίρομαι όμως που μπορώ να πω ότι πολλοί υπάλληλοι ε, πολύ ευχαρίστως βοηθούν τους επιβατές. Αυτή όμως είναι η καλύτερη ελπίδα των επιβατών για συνέχιση του ταξιδιού τους. Ε, δεν νομίζω όμως ότι η καλοσύνη κάποιου υπαλλήλου είναι αρκετά στη βαρύ βάση για τα δικαιώματα των επιβατών. Ευχαριστούμε κύριε Μιζολία και Σμιθ. Ο κύριος Ροντ έχει το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και το πάνελ των ομιλητών. Θέλω να θέσω πολλές ερωτήσεις, αλλά να ξεκινήσω από τον κύριο Λόκμαν. Μου φαίνεται ότι δεν πιστεύετε ότι πρέπει να επιβάλλουμε νομοθεσία για τα ενιαία εισιτήρια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχω όμως ένα παράδειγμα από τον προηγούμενο μήνα. Το κοινοβούλιο πήγε στο Στρασβούργο. Εγώ αγόρασα το εισιτήριο μου για το Στρασβούργο στο Νόιμουνστερ τη Γερμανίας. Ήταν εισιτήριο μετεπιστροφή. Δυστυχώς, ε, κατά την επιστροφή μου καθυστέρησα και έχασα το τρένο στο Στρασβούργο. Πήγα λοιπόν στο σταθμό και τους ζήτησα να μου αλλάξουν το εισιτήριο για το ΤΖΒ για την Καρσρούε για την Καρζούη και μου είπαν ότι δεν μπορούμε να ε, αγγίξουμε το εστήριό σας ε, διότι το αγοράσατε στη Γερμανία, στο Νόιμινστερ. Και ρώτησα, ωραία, και τι θα κάνω, διότι χρειαζόμουν κράτηση για το επόμενο ΤΖΒ. Ε, μου είπαν ότι δεν μπορώ να σας βοηθήσουν, ωραία. Ε, ε, ε, το ρίσκαρα, ανέβηκα στο επόμενο τρένο και έπρεπε να πληρώσω πρόστιμο. Μιλάμε ε, εδώ για επιχειρήσεις ε, κρατικές ε, πολύ ισχυρές. Τι πρέπει να γίνει. Να σας απαντήσω. Αυτό που αναφέρατε εσείς έχει να κάνει και με την κατάρτιση του προσωπικού. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα να ανέβετε στο επόμενο τρένο σε περίπτωση που χάσετε την, την ανταπόκρισή σας. Πάντως, εάν έχετε συμβόλαιο για ενιαίο εισιτήριο, θα ε, ισχύουν όλα τα δικαιώματα των επιβατών, ε, θα μπορείτε να ανέβετε στο επόμενο τρένο. Εάν όμως αγοράσετε ξεχωριστά το εισιτήριο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει στη δική σας περίπτωση, απλά το εξηγώ, ε, δεν μπορεί να περιμένει κανείς σε πλήρη εγγύηση, εκτός εάν υπάρχει εμπορική συμφωνία ανάμεσα στις εταιρείε να δεχτούν την κατάσταση σε περίπτωση καθυστερήσεων. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραία, σας ευχαριστώ. Προχωρώ στην επόμενη ερώτηση προς την κυρία Χαντάντ. Θα ήθελα να μας πείτε πιο συγκεκριμένα πόσο θέλετε να προχωρήσουμε όσον αφορά την παροχή συνδρομής προς άτομα με αναπηρίες. Θα ήθελα επίσης να απαντήσετε σε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Δεν συμφωνείτε ότι θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση εδώ εκτός εάν θέλουμε ε, το προσωπικό να έχει ανώτερη εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση. Ε, πώς θα το χειριστούμε αυτό. Η κυρία Χαντάτ. δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να έχουν όλοι τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα είναι να παρέχεται κατάρτιση και το να μπορεί να ταξιδεύει κάποιος με αναπηρίες ε, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με οποιονδήποτε στην Ευρώπη. Για παράδειγμα τώρα, για να πάρω ένα τρένο, ε, συχνά πρέπει να φύγω από την δουλειά μου, από μια διάσκεψη. Για παράδειγμα, αν έχω ε, μία δυνατότητα μόνο. Πρέπει να πάρω ένα τρένο στις 12 και 43. Δεν μπορώ να πάρω το τρένο που θα βγει νωρίτερα ή αργότερα. Ε, για παράδειγμα, πρέπει να ε, έχω κάνει ειδική κράτηση ώστε να έρθει κάποιος να μου ε, ξεκλειδώσει την ράμπα για να μπορέσω να μπω στο τρένο. Δεν μιλάμε για ε, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί να κάνει κάθε υπάλληλο στο στο σιδηρομικό σταθμό. Αν μπορεί να το κάνει εμένα βοηθό μου, θα μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε δουλεύει στο σταθμό. Ωραία, σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κράμερ, έχετε πέντε λεπτά. Καταρχήν ε, να πω ε, προς τον ε, κύριο Λόχμαν το 50% θέλουν αυτό το, τη μορφή εισιτηρίου. Το εξηγήσατε αλλά αρνείστε ότι όλα αυτά είναι δεσμευτικά. Γιατί όμως πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι ήδη εξήγησα ότι δεν είναι ότι είμαστε κατά της αρχής. Εμείς ε, διαφωνούμε με το να υπάρχει δέσμευση για ένα μόνο μέσο, το οποίο αποκαλείται τρένο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, παραδείγματος χάρη, ε, στην αεροπλοεία. Εγώ λέω ότι αν θέλει κανείς ότι πρέπει μόνο να ζυγίζει τα δικαιώματα των πελατών και τις εμπορικές ελευθερίες ε, των εταιριών. Βεβαίως ε, ο στόχος είναι να προσελκυστούν ως το δυνατόν περισσότεροι πελάτες. Εντάξει, τότε θα πρέπει να αγωνιστείτε έτσι ώστε όλα αυτά που μας λέτε να καταστούν δεσμευτικά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση προς τον κύριο Σμιτ. Τελικά, αν υπάρχει γενικά έτσι μια τέτοια δεσμευτική συμφωνία, πιστεύετε ότι ο αριθμό των επιβατών θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Ποια είναι η δική σας άποψη. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει δύο ειδών επιπτώσεις. Αυτοί αυτη δηλαδη που ανησυχούν προφανώς θα έχουν την εμπιστοσύνη, θα νιώθουν ότι θα αποζημιωθούν. Υπάρχουν άλλοι όμως ε, πιβάτες ε, ε, που δεν το σκέφτονται και πάνε στην κολονία και τους λένε να πληρώσουν 500 ευρώ. Αυτοί δεν θα ξαναχρησιμοποιήσουν το τρένο και θα πούνε στους φίλους τους την κακή τους εμπειρία και αυτοί θα το πούνε και παρακάτω. Εάν λοιπόν θέλουμε να επεκταθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε κατά νου. Και να πω κάτι για την αεροπλοεία. Κάποιος μου είπε ότι αν στο Βέλγιο υπήρχαν περισσότεροι σιδηροδρομικοί αστυνομικοί σταθμοί ε, θα υπήρχαν και λιγότερα αεροδρόμια. Λονδίνο, Πράγα, υπάρχει μια εταιρεία που με πάει με ένα εισιτήριο. Ε, γιατί να πάμε το τρένο όπου χρειάζομαι τουλάχιστον τρία εισιτήρια. Υπάρχουν εκεί πολλοί σταθμοί και οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι ε, να αλλάζουν συνεχώς τρένα. Αυτό, αυτές οι αλλαγές γίνονται πολύ περισσότερο από ό,τι στην αεροπλοεία. Εάν λοιπόν τελικά θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ε, σειρωμικούς ε, φορείς να έχουν ε, τη δική τους πολιτική πρέπει να βρούμε κάποια συμφωνία να έχουμε ένα σύστημα πολίσεων που να επιτρέπει ένα ταξίδι να το κάνει κανείς με μία συναλλαγή Όσο λοιπόν υπάρχει το δικαίωμα του να υπάρχει ένα ταξίδι που να είναι κανείς εξασφαλισμένος ε, νομίζω ότι αυτό για τους επιβάτες θα είναι πολύ ικανοποιητικό. Όσο όταν, όταν μιλήσατε για την ε, force majeure, για την ε, έκτακτη περίπτωση αυτό οι αεροπορικές εταιρείε το χρησιμοποιούν συνεχώς, αναγκαζόμαστε να καταθέσουμε αγωγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,3 εκατομμύρια αγωγές θα υπάρχουν ανακράτως μέλος σε 15 ε, κράτη-μέλη. Εσείς γιατί αρνείστε να εγκριθεί αυτό το θέμα της ανωτέρας βίας. Αυτό το κάνουν οι αεροπορικές εταιρείε και στην Ιαπωνία, όπου όλα είναι στην ώρα τους, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς γιατί το απορρίπτετε αυτή την έννοια της ανωτέρας βίας, της ανώτερης βίας. Κοιτάξτε, νομίζω, αν δει κανεί το κόστος, νομίζω ο μόνος τρόπος για να βελτιωθούν οι σιδηρόδρομοι είναι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 Κοιτάξτε, ακόμα και η Επιτροπή είναι επιφυλακτική σε μια έντονη διατύπωση. Ε, γιατί αν τελικά όλοι πάνε στα δικαστήρια ε, θα είναι ατελείωτος ο αριθμός των αγωγών ε, και η δική μου εμπειρία είναι ότι μετά από 1,5 χρόνο δεν γίνεται τίποτα και θα έχετε εξοικονομήσει και χρήματα. Εμείς όμως θέλουμε τα τρένα να είναι στην ώρα τους και να μην δημιουργείται κανένα είδους πρόβλημα, να μην υπάρχουν αυτές οι αγωγές. Ich denke, das, Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε τώρα στο τέλος και κατ' ουσίαν αυτό ευχόμεθα, το επιθυμούμε. Αν δούμε λιγάκι τι γίνεται στην ε, Ιαπωνία, ε, ένα τρένο, αν αργήσει, αυτό γίνεται είδηση στα εφημερίδες. Αν το κάναμε εμείς αυτό στην Ευρώπη, θα έπρεπε κάθε μέρα να έχουμε τόμους αντί για εφημερίδες. Αυτή είναι η διαφορά. Έχω πάει πολλές φορές στην Ιαπωνία ε, και λένε όλοι ότι η Ιαπωνία είναι μια ειδική περίπτωση. Ε, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί ξέρετε τι, στην Ιαπωνία η νοοτροπία είναι εξή. Ο πελάτης είναι βασιλιάς, το σημαντικότερο. Παντού ισχύει αυτό. Και πελάτης τι σημαίνει. μπορεί να θέλω μια υπηρεσία να παρέχεται αλλά με τον καλύτερο τρόπο ε, και αν αυτό περάσει σε όλα τα μέλη της αλυσίδας νομίζω ότι τότε καταλήγουμε σε μια πολύ καλή υπηρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό τον γύρο των ερωτήσεων. Τώρα μένουμε στο δεύτερο γύρο και επειδή πρόκειται για μη σκιώδης, έχετε δύο λεπτά, γιατί είσαστε πολύ. Ο κύριος Κορ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα κάνω έτσι μία λιγάκι προβοκατόρικη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, αυτή η οδηγία τελικά ε, είναι ικανοποιητική, δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί. Ε, γιατί πριν από λίγο καιρό μιλήσαμε για τις ε, πολύτροπες μεταφορές. Εσείς πιστεύετε να υπάρχουν ενιαία εισιτήρια ή μας θα πρέπει να τα σκεφτούμε λιγάκι διαφορετικά, δηλαδή να δούμε και τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Να το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ να απαντήσετε. Αξιότιμα κύριε Βουλευτά, ε, πράγματι ε, Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα για τα δικαιώματα επιβατών για διάφορα και διαφορετικά μέσα μεταφοράς. Έχουμε καταθέσει ήδη μία πρόταση ε, για τα δικαιώματα επιβατών που χρησιμοποιούν τρένο και αεροπλάνο. Όμως ε, το Συμβούλιο ε, δεν προχώρησε αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αναθέσουμε μία μελέτη για το κατά πόσον, να διαψωθεί κατά πόσον υπάρχουν τέτοια επιχειρηματικά μοντέλα και κατά πόσον σε αυτό το πολυμορφικό και πολυτροπικό πλαίσιο ε, πρέπει να υπάρχει και να εκδοχή των δικαιωμάτων των επιβατών. Τώρα τι κάνουμε, συγκρίνουμε τις μελέτες και υπολογίζουμε ε, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 να έχουμε τα πορίσματα των μελετών. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, να σας πω ότι σε έναν άλλο τομέα που αφορά στην ε, κατεξουσιοδότηση πράξη για πολυμορφικές ε, μεταφορές. Η πράξη αυτή δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβρη του 2017 και εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί βάση, δηλαδή να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και με βάση τα δεδομένα νομίζω ότι μπορεί κανείς ε, να ε, καταλήξει και σε πολυμορφικά ταξίδια. Αυτό όμως έχει σχέση και με την ενομέρωση. Μπας περιπτώσει προσπαθούμε το θέμα να το εξετάσουμε από διάφορες ε, πτυχές. Πάντως μας ενδιαφέρει και σας λέω θα ασχοληθούμε με το θέμα ε, διότι καθότι υπάρχει όλο και περισσότερη ψηφιοποίηση το πρόβλημα που θέσατε θα τίθεται όλο και περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρικέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Λόχμαν. Μιλήσαμε για το ενιαίο εισιτήριο και νομίζω ότι πριν από το ενιαίο εισιτήριο υπάρχουν θέματα επικοινωνία, επικοινωνίας στον εμπορικό τομέα, ωράρια και ε, τιμές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ισχύσει αυτό που ισχύει και στον τομέα των αερομεταφορών, δηλαδή να μπορεί ο επιβάτης να συγκρίνει τις τιμές από τις διάφορες επιχειρήσεις. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, Λόχμαν. Δεν ξέρω κατά πόσο κατανόησα την ερώτηση. Μιλάτε για εναρμόνιση τιμολόγησης. Ε, δεν είναι και τόσο απλό γιατί υπάρχει εμπορική ελευθερία να ορίσουν επιχειρήσεις τιμές όπως το επιθυμούν. Η ερώτησή μου είναι θα μπορούσε να ήταν ε, υποχρεωτική η συνεννόηση των επιχειρήσεων ως προς την τιμολόγηση και τα ωράρια, έτσι ώστε να μπορεί ο επιβάτης να συγκρίνει ωράρια και τιμές. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αυτό ακριβώς προωθούμε Γι' αυτό ε, ακριβώς μίλησα και με το ενιαίο ιστήριο, να υπάρχουν δηλαδή ε, διεπιφάνειες, ε, interfaces, για να μπορεί κανείς να ορίσει την τιμή, τα ωράρια και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό ε, θα τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό και θα συμβαδίζει με τον κανονισμό με βάση τις εμπορικές συμφωνίες των συμμετεχόντων. Άρα οι επιχειρήσεις ε, θα το κάνουν τη στιγμή που υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων. Δεύτερη ε, ερώτηση προς τον κύριο Κίντορ. Είναι δύσκολο να λάβουμε υπόψη ε, τις υπεραστικές μεταφορές με τις μακρές διαδρομές. Ε, δυστυχώς πολλές φορές δεν υποβάλλει κανείς αίτηση αποζημίωσης γιατί είτε δεν γνωρίζει είτε θεωρεί ότι η αποζημίωση είναι ελάχιστη. 2, 5, 10 ευρώ. Τι θα λέγατε να υπάρχει μία γραμμή επιβάτη όπως ισχύει με τους λογαριασμούς Miles έτσι ώστε να υπάρχει αποζημίωση η οποία να ε, χορηγείται σε ετήσια βάση. Δεν θα ήταν ε, δυνατό να υπάρχει μια κάρτα ετήσιας ε, αποζημίωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, πράγματι αλλά στην εκτέλεση χωλένει. Θα πρέπει να δούμε πώς οι επιχειρήσεις θα προβούν σε αυτή τη σύσταση. Καταρχήν, σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ εθνικών σιδηροδρομικών φορέων, που είναι όλο ένα και περισσότερα, αλλά νομίζω ότι στις αστικές μεταφορές ε, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο γιατί Πρόκειται για φτηνά εισιτήρια. Αυτό όμως που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι οι συνδρομητές που έχουν ετήσια συνδρομή, μηνιαία. Θα πρέπει δηλαδή να τους αποδοθεί η αποζημίωση ανάλογα με τις καθυστερήσεις τη στιγμή που υπάρχει, θα υπάρχει διαφάνεια. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Έχω. Το 2012 ήμουν εισηγητής σχετικά με τα ενιαία πρότυπα στους διάφορους τρόπους μεταφορών. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τι ιδιαιτερότητε του κάθε είδου μεταφορών, ε, εναρμόνιση ναι, αλλά μέχρι κάποιο σημείο. Να ρωτήσω λοιπόν πρώτον τον κύριο Λόχμαν. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πιστεύετε ότι πηγαίνει σε σωστή κατεύθυνση, πιστεύετε ότι ε, αποτελεί βήμα κατά του αθέμητου ανταγωνισμού που έχετε δει μέχρι, μέχρι τώρα. Επί της αρχής ε, ναι, θα πω ότι η πρόταση πράγματι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, προσπαθεί να εξαλείψει τις διαφορές ανάμεσα στους διάφορους ε, τρόπους μεταφορών. Θα μπορούσε βέβαια να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, για παράδειγμα να ισχύουν ε, οι ίδιες αρχές για τα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να δούμε αναθεώρηση των δικαιωμάτων επιβατών για όλα τα είδη μεταφορών ταυτόχρονα. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν ε, θα μπορέσουμε να εξετάσουμε επαρκώς το θέμα. Τον ε, Πολωνό εμπειρογνώμονα θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής. Ε, τονίσατε την ισορροπία. Αναφερθήκατε στα διάφορα πρότυπα, στα διάφορα κράτη-μέλη και μας προειδοποίησατε να μην υπερβάλλουμε στην πρόταση αυτή. Πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία αυτή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και για τα 27 κράτη-μέλη. Όσον αφορά την εξέβρεση της σωστής ισορροπίας, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία όσον αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών. Για παράδειγμα, στους σιδηροδρόμους εφαρμόζουμε κάποιους κανόνες για να υπάρχει διαφάνεια όμως και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και για τις οδικές μεταφορές, ε, τις θαλάσσιες μεταφορές ε, ή τις αεροπορικές μεταφορές. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει παρόμοια ρύθμιση. Να εφαρμόζονται, να γίνονται σεβαστά τα ε, δικαιώματα των επιβατών και σε αυτά τα είδη μεταφορών. Δεν ξέρω αν αυτό απαντά στην ερώτησή σας. Μία πολύ σύντομη τελευταία ερώτηση. προς ε, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Επιβατών. Αναφέρατε ότι δεν παρέχεται επαρκής ε, πληροφόρηση και όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής. Θεωρείτε επαρκή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα δικαιώματα προσφυγής. Προς ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας. Αφήνω τον συνάδελφο να απαντήσει και θα συμπληρώσω αν χρειάζεται. Αν κατάλαβα σωστά, η ερώτηση έχει να κάνει με τις δυνατότητες αποζημίωσης και αν είναι επαρκείς οι κανόνες. Καλά κατάλαβα την ερώτησή σας. οι επιβάτες παραπονιούνται κυρίως ότι δεν μπορούν ε, να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά τις δυνατότητες προσφυγής. Ε, Ο κύριος Σμέλτερς, ευχαριστώ πολύ. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βλέπω διάφορες προτάσεις με καλές προθέσεις για βελτίωση των δυνατότητων προσφυγής των επιβατών, την καλύτερη παροχή πληροφοριών προς τους επιβάτες. Εγώ όμως θα ήθελα να αναφέρω μια συγκεκριμένη ανησυχία. Πριν από περίπου ένα χρόνο, έθεσα το θέμα μέτρησης των καθυστερήσεων. Πώς μετράμε πόσο, πόση είναι η καθυστέρηση. Δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε με ενιαίο τρόπο τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρώπη εάν δεν έχουμε ενιαίο τρόπο υπολογισμού της καθυστέρησης. Για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη εφαρμόζουν το ε, κανόνα για τρία λεπτά, άλλα για δέκα λεπτά. Κάποια κρατημέλη υπολογίζουν την καθυστέρηση στη, στον τελικό προορισμό, άλλα υπολογίζουν την καθυστέρηση και στους ενδιάμεσους σταθμούς. Ε, κάποιοι υπολογίζουν με βάση αριθμό επιβατών. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι διάφοροι τρόποι υπολογισμού των καθυστερήσεων και δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία από χώρα σε χώρα. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να δώσουμε καλύτερες πληροφορίες στους επιβάτες σχετικά με τις καθυστερήσεις. Ε, στην χώρα μου υποτίθεται ότι πρέπει να δημοσιεύονται τρεις φορές τη μέρα ε, τα στοιχεία περί καθυστερήσεων, αλλά δεν έχουμε σύστημα συγκρίσιμο. Εάν είχαμε ένα πρότυπο σύστημα, αυτό θα ήταν χρήσιμο για τους επιβάτες, διότι έτσι θα μπορούσαν να συγκρίνουν στοιχεία των διαφόρων εταιριών. Οι ομιλητές μας ε, λοιπόν ε, τι γνώμη έχουν ε, όσον αφορά τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος για τον υπολογισμό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σμίθ ή ο πρόσωπος της Ένωσης των Επιβατών θα μπορούσαν να απαντήσουν. Νομίζω ότι πρέπει να επιταχύνεται γιατί θα πρέπει να φύγουν και οι ενδιαφερόμενοι πάνελιστ. Σε ποιον απευθύνεται την ερώτηση. Uh, ε, ο κύριος Μέλντερς ναι, νομίζω πράγματι ότι το θέμα της αναχώρησης στην ώρα του ε, των τρένων είναι πολύ σημαντικό θέμα και ε, όπως υπόθηκε αναγκάσαμε την Ινφραμπελ να μας δώσει καλύτερα στατιστικά στοιχεία. Αύριο θα συζητήσουμε εις βάθος μαζί του το θέμα αυτό. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως, διότι συνεχώς αυτό συζητιέται και εσωτερικά στις οργανώσεις μας. Κάθε χώρα έχει δικούς τους κανόνες και, και δικό της τρόπο υπολογισμού. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού, διότι στις συζητήσεις που είχαμε με την SNCB και την Infrabel σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των καθυστερήσεων, τελικά μας εξήγησαν τον τρόπο που το υπολογίζουν, αλλά μετά από πολλές προσπάθειες, διότι δεν ήθελαν να είναι πολύ διαφανείς στο θέμα αυτό. Πρώτη το πρώτο μας μήνυμα λοιπόν είναι να είστε διαφανείς, να παρέχετε πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα στοιχεία. Εξηγήστε μας πώς το υπολογίζετε, διότι όπως είπατε αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να, είναι, να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Ευχαριστώ ο κύριος Βιμ Φαντεκάμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμένα στη συζήτηση αυτή μου κάνει εντύπωση ότι ξεχνάμε ότι οι σιδηρόδρομοι είναι ο τομέας μεταφορών που λαμβάνει τις περισσότερες ενισχύσεις. Ε, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο αυτό που υπόθηκε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τον οδικό τομέα. Μπορούμε, διότι είναι ο τομέας που λαμβάνει τις περισσότερες ενισχύσεις. Ένα υποχρεωτικό σύστημα λοιπόν για ενιαία εισιτήρια δεν ε, θα είναι χρήσιμο και εφικτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς αυτό το εργαλείο για να αναγκάσουμε να υπάρξει διασυνοριακή συνεργασία. Απογοητεύτηκα πολύ από αυτά που άκουσα από τον Πολωνό ομιλητή, διότι επιλέγει τις επενδύσεις εις βάρος ε, των ε, επιβατών, αν κατάλαβα καλά. Εδώ Ίσως η ερώτηση είναι προς τον κύριο Ολζέσκι. Α, όχι, δεν είναι θέμα ερώτησης. E, Αν θέλετε μπορώ να απαντήσω. Αν αυτό είναι επιθυμητό. Εγώ είμαι υπέρ των επενδύσεων ε, για τους ε, επιβάτες. Η PKP, η επιχείρησή μας, αυτή τη στιγμή προβαίνει σε ένα σχέδιο επενδύσεων για τους σταθμούς, έτσι ώστε να έχουμε όλες τις τεχνολογίες εχμής για τους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα. Θέλουμε να άρουμε τα ε, αρχιτεκτονικά προσκόμματα και θα θέλαμε να επενδύσουμε και στο τροχαίο υλικό έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικά μία ε, πλήρης επένδυση Η ερώτησή μου προς τον κύριο Λόχμαν. Μπορείτε να την επαναλάβετε, παρακαλώ. Euh, euh, Το σχόλιο άκουσα, αλλά δεν επρόκειτο για ερώτηση. Ε, κύριε Λόχμαν, ο κύριος Λόχμαν την κατάλαβε πάντως. Θα ήθελα να ακούσω και την απάντησή του. Εντάξει. Εκείνος άκουσε την ερώτηση, Λόχμαν. Ναι, πράγματι ο κύριος Λόχμαν κατάλαβε την ερώτηση ε, και δεν συμφωνεί με το θέμα, με την δήλωσή σας ότι λαμβάνει τις περισσότερες ενισχύσεις ο συνδρομικός τομέας. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις ε, ε, ενισχύσεις και τις επενδύσεις στο οδικό δίκτυο. Μπορούμε όμως μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες, αλλά όπου υπάρχει εμπορική ελευθερία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ε, κανόνα. Ε, ε, μιλάμε εδώ για δύο, διαφορετικά, δύο διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Η κυρία Αρνότου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους παρεμβαίνοντες. Εγώ έχω μία ιδιάζουσα ερώτηση προς τον κύριο που αντικαθιστά τον κύριο Γκαζού. Άκουσα για τα δικαιώματα επιβατών, αλλά νομίζω ότι το πρώτο δικαίωμα είναι η ασφάλειά τους κατά την ε, μετάβαση την διαδρομή τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον. Και επίσης σιδηροδρομικές υπηρεσίες, σωστές, ακριβείς και ούτω καθεξής και ασφαλείς βεβαίως, πρωτίστως. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι μείωση του προσωπικού σιδηροδρόμων και πολλές φορές υπάρχουν και λαιλασίες Πέρυσι η γαλλική υπηρεσία, μια γαλλική υπηρεσία ε, ότι το 40% των επιβατών θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλής και το 37% των πράξεων βίας, ιδιαίτερα κατά των ε, γυναικών, ε, αφορά τους σιδηροδρόμους. 56% έναντι 26% ανδρών. Πολλοί μιλάνε για βαγόνια ε, που θα πηγαίνουν μόνο γυναίκες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ουσιώδες πρόβλημα. Πώς μπορεί να επιληθεί και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την Επιτροπή για αυτό το θέμα που είναι πολύ ε, φλέγον. Κιντόρ, θα πρέπει να σταθούμε στην ασφάλεια πρωτίστως. Θεωρώ ότι η σιδηρόδρομη είναι το πιο ασφαλές ε, μέσον ως προς τα δυστυχήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς. Εμείς θεωρούμε στην Ομοσπονδία Χριστών ότι η σιδηρόδρομη είναι ένα από τα πιο ασφαλή μέσα. Ως προς την ασφάλεια κινήσεων βλέπουμε ότι μία στις δύο γυναίκες είναι θύμα κάποιας μορφής βίας και γι' αυτό προβήκαμε σε μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης γιατί το θέμα αφορά τους χρήστες, αλλά δεν πρέπει οι χρήστες να αναλαμβάνουν την ασφάλειά τους. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να δράσουν, αστυνομία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Η κυρία Συναλόβα για δύο λεπτά. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της μεταφοράς των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα. Στο Intergroup μιλήσαμε, θα μιλήσουμε για το θέμα την επόμενη Τετάρτη προς τον κύριο Λόχμαν θα ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση. Ακούσαμε για τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της ανάγκης ε, του να κλείνει το εισιτήριο κανείς ε, εγκαίρος online όπως είπε και η κυρία Χαντάντε, γιατί υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφοροποιήσεις. Είναι θέμα οργάνωσης, εξοπλισμού, κακής θέλησης. Οι διαφορές οφείλονται κυρίως στο ότι τα είδη υπηρεσιών δεν είναι όμοια στις ε, χώρες που αναφέρατε, όπου είναι υψηλή η πυκνότητα της κυκλοφορίας, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι πολύ διαφορετικές από σε περίπτωση που είναι πολύ αραιή η κυκλοφορία ή έχουμε σταθμούς με προσωπικό και χωρίς. Ε, θα πρέπει λοιπόν στην ε, περίπτωση των ε, ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα δεν έχουμε πρόβλημα να μειωθεί ο χρόνος προειδοποίησης ή να παρέχονται υπηρεσίες που να μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς χωρίς επιπλέον βοήθεια. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Χαντάτη έχει να απαντήσει. Νομίζω ότι πολύ συχνά είναι θέμα καλής βούλησης, διότι συχνά ήδη υπάρχει ο εξοπλισμός. Δεν θέλουμε κάτι υπερβολικό. Θέλουμε απλά πρόσβαση στις σιδηροδρομικές μεταφορές όπως έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ε, όταν μιλάμε για κατάρτιση και εσείς μου λέτε ότι όχι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ευιστοτοποιήσουμε ε, όλους σχετικά με τις δυνατότητες που έχουμε. Ε, για πρόσβαση, διότι πολύ συχνά υπάρχει εκεί ο εξοπλισμός, απλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται κιόλας. Η κυρία Άντερσον για δύο λεπτά, τελευταία παρεμβαίνουσα. Σας ευχαριστώ που μου ξανατείνετε το λόγο. Οι σοσιαλιστές έχουν αναλάβει αυτήν την ε, έκθεση στην ΤΡΑΝ, αλλά είμαι και σκιώδης εισηγητής ε, ε, για την έκθεση αυτή σε άλλη επιτροπή. Και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα άρθρα 7 και 12 της συνθήκης για να διασφαλίσετε την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και για να διασφαλίσετε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Και επίσης όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν συμφωνείτε ότι οι συνδρομικοί φορεί θα πρέπει να αναγκαστούν να αναλάβουν ε, ε, να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα της επίλυσης διαφορών ε, χωρίς να θίγονται άλλα δικαιώματα των καταναλωτών. Αν δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν την εναλλακτική επίλυση διαφορών οι συνδρομικοί φορείς, δεν θα προχωρήσουμε πολύ όσον αφορά την επιβολή των των νόμων και τον ε, σεβασμό ε, των δικαιωμάτων των επιβατών. Ε, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι προσπαθούμε να πετύχουμε προόδο και να έχουμε εναλλακτική και επιγραμμική επίλυση διαφορών. Μέχρι τώρα όμως δεν ε, έχει καταστεί υποχρεωτική όπως προτείνετε εσείς αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή Ε, έχουμε συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και συζητάμε αυτές τις νέες μεθόδους επίλυσης διαφορών, ε, τις εναλλακτικές και τις επιγραμμικές, με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, διότι διαπιστώσαμε ότι δεν είναι όλες ενήμερες σχετικά με ε, τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν. Θέλουμε επίσης να δίδονται συστάσεις για την χρήση αυτών των μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Είναι όμως σχετικά νέα εργαλεία και θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές οδηγίες. Οι συνάδελφοί μας ε, της νομικής υπηρεσίας εξετάζουν το θέμα και πράγματι έχετε απόλυτο δίκιο Περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα. Πάντως αυτή τη στιγμή μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε στην πράξη να εφαρμόσουμε τους κανόνες. Άλλωστε είδατε ότι μόλις επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός ε, για την ε, προστασία των καταναλωτών και ότι όλοι οι κανονισμοί για τις μεταφορές, ε, δηλαδή και αυτός για τους σιδηροδρόμους και ε, για τις αεροπορικές μεταφορές και τις οδικές μεταφορές ε, καλύπτονται. Αυτό πάντως που προτείνατε μπορεί να είναι κάποιο επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή θα παραμείνουμε σε αυτά που έχουμε και θα προσπαθήσουμε πρώτα να εφαρμόσουμε αυτούς τους σχετικά νέους κανόνες. Ευχαριστούμε πολύ για την τελευταία παρέμβαση. Θα ήθελα ο Ισμαήλ Ερτούγκ Α, όχι, η κυρία Άντερσον θα συνοψίσει. κυρία Άντερσον, ξανά ελάτε εδώ στο προσκήνιο. Ναι, με βοήθησε αυτή η απάντηση, αλλά διαφωνώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο... Δεν είμαστε πια στη συζήτηση. Θα πρέπει να συνοψίσετε στη θέση του εισηγητή πολύ χρήσιμη η συζήτηση που θίγει ορισμένα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ως προς τη, τα θέματα που αφορούν τις αναπηρίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κυρίως έντοτε υπάρχει μια νέα νομοθεσία περί προσβασιμότητας. Πραγματικά πιστεύω ότι από πλευράς ε, των φορέων. Συμφωνώ με τον Δήμο ότι όλα αυτά που συνέβησαν είναι απογοήτευση. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο θετικοί γιατί νομίζω ότι ε, είναι σημαντικό οι επιβάτες να νιώθουν εμπιστοσύνη όταν ταξιδεύουν με το τρένο. Όλοι θέλουν το τρένο να ταξιδεύει γρήγορα και αν έχουμε τόσο περιορισμένη άποψη δεν θα τα καταφέρουμε. Δικαιώματα βεβαίως των επιβατών σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές. Ε, αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Άντερσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονες για το χρόνο τους, αλλά το θέμα μόλις έχει ανοίξει. Άρα Ελπίζω να έχουμε και άλλες ανταλλαγές απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην Επιτροπή μας και να σας χειροκροτήσουμε. Et vous pouvez aussi applaudir mon bras, mon qui a été très très sage, il a été très attentif, vous avez vu. Hein Et en tout cas, j'espère que tu... Ελπίζω να ε, βρεις το χρόνο να ανακαλύψει το κοινοβούλιο, λέει η πρόεδρος στον φιλαράκο της δίπλα και περνάμε στο επόμενο θέμα της Ελβετίας, της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών. Ah, C'était Euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10. La délégation suisse, venez me rejoindre. Η ελβετική αντιπροσωπεία να έρθει εδώ.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

Merci. Nous continuons notre échange de vues avec, on a l'honneur d'avoir dans notre délégation, Monsieur l'ambassadeur. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ μαζί μας, γιατί θα μας ε, μιλήσετε για την ε, ελβετική οπτική των μεταφορών, ο κύριος Φουγκλιστάρελερ είναι υπεύθυνος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών και μας ενδιαφέρει οι διατροπικές μεταφορές. Έχετε 10 λεπτά για να μας μιλήσετε για την πείρα σας και στη συνέχεια θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα μπορέσω να μείνω μέχρι τέλους. Ο κύριος Ρικέ θα με αντικαταστήσει, αλλά θα σας δω στο εγγύης μέλλον. Μπορούμε να αρχίσουμε. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά για αυτές τις διατροπικές μεταφορές. Να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελβετία. Madame la Présidente, merci beaucoup pour cette introduction τηρήσω το ωράριο όπως κάνουν όλοι οι Ελβετοί. Θα μιλήσω αγγλικά, νομίζω ότι είναι η καλύτερη, ε, είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω, γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε απευθείας αγγλικά. Όπως ξέρετε, η ελβετική πολιτική είναι η Για μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα από τους δρόμους ε, στα τρένα με φιλική ε, προς το περιβάλλον πολιτική και προσπαθούμε και να ενταχθούμε και στην ευρωπαϊκή πολιτική, βεβαίως με την ευθύνη τη δική μας της ε, Ελβετίας. Η πολιτική αυτή η μεταφορά από ένα μέσο σε άλλο, εκεί ε, χρησιμοποιούμε τρία μέτρα. Πρώτον, νέα υποδομή, θα μιλήσω επ' αυτού. Το δεύτερο είναι η απελευθέρωση στον ε, συνδροδομικό τομέα και σήμερα θα σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα για τα τέλη βαρέων ε, οχημάτων. Αυτό είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία ε, για την ε, αλλαγή από ένα μέσο σε άλλο. Όσον αφορά την υποδομή. Πέρυσι ε, είχαμε ε, το, τη σύραγγα στο Κοτάρ που άνοιξε. Είναι το, η μεγαλύτερη σύραγγα που υπάρχει στον κόσμο και το 2020 ε, θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο άξονας και με το τρίτο με την τρίτη σύρακα και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στην Ελβετία και την Ολβετία, Ολλανδία και Ελβετία. Θα έχουμε ε, και ε, μεγάλα φορτηγά που θα μπορούν να διασχίζουν τη σύραγγα. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία Δηλαδή ε, δίνουμε πλέον τη δυνατότητα ε, στους σιδηρόδρομους να είναι πιο αποτελεσματικοί. Βέβαια δεν αρκεί αυτό ως υποδομή. Είναι όλα αυτά ε, απολύτως απαραίτητο είναι να χρησιμοποιεί κανείς και τη σωστή φορολογία. Γι' αυτό και θα έχουμε τα τέλη βαρέων οχημάτων που τα εισαγάγαμε το 2001 με βάση την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Ε, καλύπτονται έτσι οι εξωτερικές δαπάνες ε, τα τέλη ε, καλύπτουν όλα τα φορτηγά των 3,5 τόνων και ο υπολογισμός γίνεται με βάση το μέγιστο βάρος, την απόσταση και τις εκπομπές. Ε, το τέλος αυτό είναι ε, ένα τέλος που αφορά τον καταναλωτή. Κάθε χρόνο μιλάμε 1,4 δις που εισπράττονται και το 75% του τέλους προέρχεται από ελβετικά φορτηγά. Ε, τα τρία τέταρτα πληρώνονται από τα ελβετικά φορτηγά που μετακινούνται στην ε, Ελβετία και το ένα τέταρτο από τα transit φορτηγά. Ε, τα δύο τρίτα καταβάλλονται στην Ομοσπονδία η οποία χρηματοδοτεί τα μεγάλα έργα όπως τη σύραγγα στο Κοτάρ. Το 1 τρίτο των εσόδων καταβάλλεται στα καντόνια ε, και αυτοί χρησιμοποιούν τα χρήματα, τα καντόνια χρησιμοποιούν τα χρήματα για υποδομές ε, που δεν μπορούν να καλύψουν διαφορετικά. Βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα των τριών κατηγοριών τελών, ε, διοδίων, έχουμε την ε, ε, κατηγορία Euro 6 που είναι 30% κάτω από την πρώτη κατηγορία και βλέπετε όλο αυτό πολλαπλασιάζεται χιλιομετρικά και με το βάρος. Έχουμε λοιπόν διαφορετική τιμολόγηση. Στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ορίσει 325 ελβετικά για τα 300 χιλιόμετρα από το βορρά προς το νότο. Αυτό είναι το ανώτατο ποσό διοδίων και με βάση την ελβετική νομοθεσία έχουμε το μέγιστο εξωτερικό κόστος όπου εκεί ε, μπορούμε να πάμε πιο πάνω αλλά πρέπει να σεβόμαστε τη συμφωνία και την ελβετική νομοθεσία και γι' αυτό είμαστε πολύ κοντά στο μέγιστο ποσό. Όσον αφορά τώρα αυτά τα νέα μέτρα ε, βρισκόμαστε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το 99 είχαμε ως όριο τους 80 τόνους. 3 τόνοι ε, μεταφέρθηκαν με 1,3 εκατομμύρια φορτηγά. Ε, το 2016 είχαμε πολύ λιγότερα φορτηγά τα οποία μετέφεραν 11,7 τόνους και βλέπετε ότι ο μέσος όρος αυξήθηκε σε αυτή την περίοδο από 6,3 τόνους σε 12 τόνους ε, δηλαδή κατ' ουσίαν είχαμε διπλασιασμό σε λίγα μόνα χρόνια. Ε, τα διόδια αυτά συμβάλλουν και στην συνεχή ανανέωση του στόλου των οχημάτων. Είχαμε το 1, το 2001 το 82% με, 0, με 0,1 ή 0,2 το 17 είχαμε μόνο 1% τέτοιων οχημάτων. Το 92% όλων των υπηρεσιών μεταφέρονται με ε, φορτηγά Euro 5 ή Euro 6. Μελετήσαμε τις επιπτώσεις ε, από αυτά τα διόδια και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η αύξηση μόνο 0,1% για κάθε καταναλωτή αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε και παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας και το κόστος δεν μπορούσε να μετακυλιστεί όλος τους ε, καταναλωτές. Ε, το κόστος της μεταφοράς ήταν μόνο ένα μικρό ποσοστό του τελικού προϊόντος. Τέλος, βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια ότι έχουμε μαζική μείωση της, ε, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ε, το μπλε χρώμα που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια από το 2004 μέχρι το 2016 Μειώθηκαν οι εκπομπές κατά περίπου 80% και σήμερα τα βαριά φορτηγά πλέον ε, δεν είναι το ε, πιο ρηπογόνο μέσο μεταφοράς. Ο λόγος είναι βέβαια ότι έχουμε καλύτερη τεχνολογία, υψηλότερη αποτελεσματικότητα και επίσης λιγότερες μεταφορές στην ε, ε, μεταφορά στην επιλογή άλλων μέσων βλέπουμε μία μείωση ε, από το 2000 παλαιότερα είχαμε τα βαρέα οχήματα που κατέβαλαν και αυτά ένα τέλος τώρα έχουμε περιοριστεί όσον αφορά την αλλαγή μέσου μεταφοράς. Το 2016 το 71% ε, των εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν με σιδηρόδρομους και μόνο 29% μέσω χερσαίων μεταφορών. Το τέλος βαρέων οχημάτων μπορεί να κριθεί ως επιτυχία. Ε, αυτό το τέλος συνέβαλε σημαντικά στην μεταφορά ε, της συγκοινωνίας πλέον προς τους σιδηρόδρομους. Έχουμε πλέον μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των χερσαίων μεταφορών ε, με την εφαρμογή της αρχής οριπένων πληρώνει. Ε, οι επιπτώσεις στις τιμές του καταναλωτή παραμένουν πολύ χαμηλές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίασή σας. Μας εξηγήσατε τι μηχανισμοί ε, σας βοηθούν να πετύχετε τους στόχους σας. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στη συζήτηση και δίνω το λόγο στην κυρία Σμιτ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ζηλεύω πρέπει να πω αυτά που άκουσα. Αλλά <laughs> η Ελβετία μάλλον είναι ο μονόφθαλμος που βασιλεύει στους τυφλούς στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει δισεκατομμύρια που προέρχονται από φορολογικά έσοδα. Αντιμετωπίζουμε όμως σημαντικά προβλήματα Βλέπουμε όμως ε, και τα στοιχεία που δείχνουν από το 1995 μέχρι σήμερα. Είχαμε αύξηση από το 6,6% στο 6,7%. Αυτό λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Βλέπουμε ότι στις μεταφορές φορτίων είναι κάπως καλύτερα τα στοιχεία, αλλά θα πρέπει να συγκρίνουμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, και την Ρωσία και εδώ βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πίσω. Οι οδικές μεταφορές και οι αεροπορικές μεταφορές τα πάνε καλύτερα από τη σιδεροδρομή. Ιδιαίτερα με ενδιέφερε αυτό που είπατε στο τέλος της παρουσίασής σας σχετικά με τα βαρέα φορτία. Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αυστρία επιθυμούμε Ε, τα τέλη να δαπανώνται για συγκεκριμένους ε, σκοπούς. Ε, εάν διαθέσουμε έτσι τα χρήματα θα μπορέσουμε να φροντίσουμε να ε, οδηγήσουν σε μεταφορά στους σιδηροδρόμους, κάτι που θα επιθυμούσαμε και για περιβαλλοντικούς λόγους. Πρώτη ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων θα πρέπει να απελευθερωθεί όπως είδαμε σε αεροπορικές μεταφορές και τις οδικές. Στην Αυστρία αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή. πόσο μάλλον εάν συγκρίνουμε με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους, τους γερμανικούς κλπ. Επίσης, τι μέλλον πιστεύετε ότι θα έχουν οι σιδηροδρόμοι σε 10 χρόνια που γνωρίζουμε ότι θα έχουμε αυτόνομη οδήγηση και μάλιστα και από φορτηγά. Και πιστεύετε ότι η Ευρώπη μπορεί να μάθει κάτι από την Ελβετία ή θεωρείτε ότι είσαστε η θεωρειτε οτι εισαστε οι εξαίρεση που ε, επιβεβαίωνε τον κανόνα 28 ε, κράτη-μέλη δεν κατάφεραν αυτά που καταφέρατε εσείς μόνοι σας. Πάντως ζηλεύουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντεκάμπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν από δύο χρόνια μαζί με τον Μιχαήλ Κράμερ επισκεφτήκαμε ε, το πέρασμα του Μπρένερ και εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό φορτηγών που περνούσαν από εκεί. Καταλαβαίνω γιατί η Ελβετία λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα. Παρόλα αυτά, γίνονται συζητήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο τούνελ Γκότχαρτ. Και το ίδιο νομίζω θα συμβεί και για το πέρασμα Μπρένερ. Εσείς λέτε ότι το τούνελ Γκότχαρτ θα είναι έτοιμο το 2020. Την πρόβλεψη αυτή που τη βασίζεται. όσον αφορά και τους δρόμους πρόσβασης. Επίσης, αν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι τα τρία τέταρτα των φορολογικών εσόδων πληρώνονται από ελβετικά φορτηγά, ενώ το ένα τέταρτο από ε, φορτηγά που περνούν από τη χώρα. Με εκπλήσει αυτή η αναλογία. Εάν έχετε γερμανικό φορτηγό που παραδίδει... Ε, που παραδίδει αγαθά στην Ελβετία ε, πάλι χρεώνεται το τέλος ε, και πώς εισπράτεται τα τέλη αυτή. Υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Ευχαριστώ. Ναι, καταρχάς, σας ευχαριστώ κύριε Φίλιπ για την παρουσίαση αυτή. Που είναι συναρπαστική για μας. Οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλώ ε, έχουν ε, φυσικά προτίμηση για ε, τις σιδηροδρομικές μεταφορές που είναι και φιλικές προς το περιβάλλον και εσείς εδώ αποτελείτε υπόδειγμα. Αναφερθήκατε και στους στόχους που έχετε, στα μέτρα που έχετε λάβει για περιορισμό του θορύβου στις σιδηροδρομικές μεταφορές και Δεν ξέρω μήπως μπορείτε να μου πείτε, διότι πιο πολύ με ενδιαφέρει. Να μάθω στην Ελβετία ε, πώς ε, ε, έχετε χρηματοδοτήσει τον εξυγχρονισμό του τροχαίου υλικού. Μας αναφέρατε την αναλογία 1 το 2 τρίτα με αυτό το earmarking που γίνεται, την ε, διάθεση των πόρων για συγκεκριμένους σκοπούς, ε, πώς εφαρμόζεται το σύστημα. Πάντως, συγχαρητήρια, διότι πράγματι αποτελείται υπόδειγμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κάμερ, ο κύριος Φουγκλιστέρ και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φίγκλιστερ και από τον κύριο Μπιουσέ γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Ε, και θα ήθελα να σας πω ότι σας ζηλεύουμε γιατί λειτουργείτε ως, σαν ελβετικό ρολόι. Ελπίζω το ίδιο να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί και εμείς χρειαζόμαστε βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να μοιάζει το σιδηροδρομικό μας δίκτυο αύριο με το δικό σας. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την εισήγησή σας. Βεβαίως είναι λυπηρό το γεγονός ότι τώρα στην αίθουσα είναι πάρα πολύ λίγοι βουλευτές η ε, Επιτροπή θα έπρεπε να εκπροσωπείται κατά 100% και όλα τα κράτη-μέλη για να δούνε όλοι ότι το θέμα δεν είναι να ε, καταθέτουμε κάποιες απόψεις ή να εκδίδουμε ανακοινώσεις. Εσείς ε, είσαστε εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν με θαυμάσιο τρόπο τη δική μας την πολιτική το να μεταφερθούν οι μεταφορές από τους δρόμους, τους σιδηρόδρομους. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν καινούριε, απλά να κάνουμε και να μιμηθούμε αυτά που κάνετε εσείς. Βασικά αυτό θα έπρεπε να το κάνουν όλα τα κράτη, αλλά ούτε καν και αυτό δεν γίνεται. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει λάθος ε, ιεράρχηση. Ε, πολύ ωραίο αυτό που είπατε, ότι τα τρία τέταρτα των εσόδων έρχονται από ελβετικά φορτηγά. Αυτό οφείλεται βέβαια ε, στο ότι έχετε διόδια τα οποία ε, καταβάλλονται από όλα τα φορτηγά των 3,5 τόνων. Δηλαδή δεν λέτε ανάλογα με το φορτηγό και ανάλογα με το ποια θα είναι διαδρομή. Παλιότερα επιβάλλονται διόδια εκεί που πάνε οι ξένοι, αλλά είπατε ε, επιβάλλονται διόδια σε όλους. Και επειδή ε, υπάρχει αυτό, υπάρχει συνεργασία και υπάρχει και ανταγωνισμός. Ε, δηλαδή στην Ελβετία καμία εταιρεία δεν θα έκανε μία διαδρομή με δέκα μόνο κυβότια. Ε, θα απευθυνόταν σε κάποιον άλλον να τα δώσει αλλού και ο άλλος θα πήγαινε την επόμενη μέρα στον πρώτο. Έτσι λοιπόν μειώνεται το κόστος ε, και ε, με βάση τα διόδια τελικά οι καταναλωτές ε, πληρώνουν μόνο 0,5% παραπάνω. Πιο φτηνή προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί καν να υπάρξει. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά άδεια φορτηγά γιατί είναι φτηνές οι διαδρομές. Για όλα αυτά που κάνετε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως υπήρξε και δημοψήφισμα, δημοψήφισμα για, για τη σύραγγα στο Κοτάρ. Ε, με την απαγόρευση παράλληλα να κατασκευάζεται και αυτοκινητόδρομος. Κάτι τέτοιο ούτε καν μπορεί κανείς ε, ε, να το σκεφτεί στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ας πούμε στη Γερμανία, στο Τύρινγκερ Βάλτ, εκεί παράλληλα κατασκευάστηκε και αυτοκινητόδρομος. Ούτε καν σκέφτηκε κανείς να εγγύεται τις μεταφορές και να είναι ευχαριστημένος με το τρένο. Για όλα αυτά λοιπόν ένα θερμότατο ευχαριστώ και εγώ σας λέω, είσαστε μια τόσο ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε να είστε, γιατί ακριβώς δεν είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω τώρα δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι από το 2020 δεν ε, θα υπάρχουν πλέον εμπορευματικές μεταφορές μέσω Ελβετίας. Τώρα το κάνει αυτό και η Γερμανία. Και κατ' ουσίαν αυτό είναι πολύ απλό να εφαρμοθεί στην Ευρώπη. Εγώ θα επιθυμούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ότι αυτό που κάνει η Ελβετία μπορούμε και εμείς να το κάνουμε από το 2020. Και επιτρέψτε μου και μια κρίσιμη παρατήρηση ε, όταν ε, δηλαδή είχαμε το πρώτο ΙΤΣΕ ε, στην Ελβετία, τότε η Ελβετία είχε πει ότι αυτό αυτό γίνεται μόνο αν πάρει κανείς και το ποδήλατό του. Και τότε είχε πει η Deutsche Bahn ότι εντάξει θα το κάνουμε αυτό για δύο χρόνια, μετά θα υπάρξει μια αξιολόγηση και θα δούμε. Και μετά από δύο χρόνια καταργήθηκε το μέτρο, αλλά η αξιολόγηση δεν έχει γίνει καν μέχρι σήμερα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε αυτό, ε, γιατί στους ε, σιδηρόδρομους ε, υπάρχει το νέο ICE να επιβάλλεται σε όλα τα τρένα να παίρνει κανείς και το ποδήλατό του. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 44 ε, εκατομμύρια ποδηλατικό τουρισμό. Είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα από τις κουραζιέρες που είναι 39 εκατομμύρια. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ. Κάθε καλό. Εσείς αγωνίζεστε για την κινητικότητα και για το κλίμα και αυτό δεν είναι αντίφαση και μας έχετε αποδείξει πώς μπορεί να γίνει. Πριν δώσω το λόγο στο κύριο Φουγκιστάλερ, θα ήθελα κι εγώ να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος. Όπως ξέρετε, ε, έγιναν πολλά δημοψηφίσματα στην Ελβετία, τέσσερα τον αριθμό και, υπήρχανε και υπήρχε και ειδική φορολόγηση η οποία έπρεπε να προχρηματοδοτηθεί. όχι μόνο από τον φόρο για τα βαρέα οχήματα. Αυτός ο φόρος ε, ορίζει την αρχή ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή σχετίζεται με την χρήση ή είναι ε, ένας καταποκοπήν φόρος. Δεύτερον, ο φόρος αυτός είναι στοχοθετημένος, αφορά ε, θέματα εσωτερικής ή εξωτερικής ανάθεσης, έργων υποδομής, ε, αντιμετώπισης της ε, ρήπανσης και ε, ούτω καθεξής. Πώς ορίζεται αυτή η στοχοθέτηση. Ο κύριος Κράμερ έχει ακόμα ένα λεπτό. Ε, ξέχασα δύο πράγματα να σας πω. Ε, μιλήσαμε για τα δικαιώματα των επιβατών. Μήπως ε, μπορείτε λιγάκι να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα δικαιώματα των επιβατών στην Ελβετία. Και το δεύτερο, να πω το εξή. η σύραγγα του Γκοτάρ συνήφθη η Συμφωνία Ολλανδία, Ελβετία, Ιταλία για 21 χρόνια. Έχει τελειώσει το η σύραγγα, αλλά όχι η παράπλευρη δρόμη. Η Γερμανία λέει ότι το 43 ε, θα είναι έτοιμη οι παράλληλη δρόμοι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Άκουσα στην Ιταλία ε, γίνονται κατασκευές, αλλά μόνο με τα δικά σας χρήματα. Το ότι δεν τηρείται η σύμβαση Μήπως σκέφτεστε να ε, καταθέσετε αγωγή κατά των κρατών, γιατί το να είναι μόνο έτοιμη σύραγα και όχι η παράπλευρη δρόμη, αυτό δεν είναι καλό για την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν μία σειρά ερωτήσεων και αφού ακούσατε όλες ε, τις φιλοφρονήσεις μας έχετε και το λόγο για να μας απαντήσετε. Σας ε, δίνω το λόγο για 10-12 λεπτά το πολύ για να απαντήσετε σε αυτή τη σειρά των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τους πολλούς επένους που άκουσα και από την κυρία Σμιτ. εάν θέλετε μεταφορά των μεταφορών στους σιδηροδρόμους ε, θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια από όλες τις πλευρές ε, και γι' αυτό στην Ελβετία ανοίξαμε πολύ νωρίς ε, αυτόν τον ανοιχτό άξονα για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Χρειάζεται και ε, κάποια πρόβλεψη για τους σιδηροδρόμους. Φυσικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό σε διάφορες χώρες. Ε, για παράδειγμα ε, χωριστή ευθύνη, υποδομές κλπ. Πάντως μπορεί η αποτελεσματικότητα να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους. Καλά θα κάνουν όμως οι χώρες να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο τρόπο για αυτές. Όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση σε 10 χρόνια προβλέπεται κάτι τέτοιο και υπάρχουν ιδέες για το λεγόμενο πλατούνινγκ να ε, συνδέονται δηλαδή οχήματα μεταξύ τους. Ε, κάτι παρόμοιο που γίνεται και στους σιδηροδρόμους που έχουμε μία μηχανή και διάφορα βαγόνια από πίσω. Ε, οι σιδηρόδρομοι είναι μέσω μαζικής μεταφοράς ε, και γι' αυτό ε, μας ενδιαφέρουν οι μεγάλοι όγκοι. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι και σε 10 χρόνια πάλι θα βρισκόμαστε μπροστά από τις οδικές μεταφορές. για μεγάλες αποστάσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η σιδηροδρομή. Ε, ναι, λέτε να μάθετε από την Ελβετία, γιατί όχι άλλωστε και εμείς μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, την διαλειτουργικότητα την υιοθετούμε, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ε, μεταφοράς αγαθών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Η Ελβετία εποφελείται από αυτές ε, τις ενιαίες προδιαγραφές αντί να πρέπει να συνεννοηθεί με κάθε ξεχωριστή χώρα ε, σχετικά με τις προδιαγραφές. Νομίζω ότι πρόκειται για διαδικασία αμοιβαία μάθησης. Πότε έχει ο ένας μια καλή ιδέα, πότε έχει ο άλλος. Και νομίζω ότι και στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ένα από τον άλλο. Πάντω, όσον αφορά του σιδηροδρόμου, είχαμε πράγματι κάποιε καλέ ιδέες. Κύριε Κράμερ και κύριε Βίμτεκάμπ, ε, αναφερθήκατε στους δρόμους πρόσβασης. Το 2020 ε, θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρόμοι στην ε, Ελβετία, από τη Βασίλεια δηλαδή, και με την Γερμανία και την Ιταλία έχουμε την συμφωνία ώστε να αυξηθεί η ικανότητα, το δυναμικό των δρόμων πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες Η Ιταλία λοιπόν ε, ε, έχει ε, προσπεράσει τους Γερμανούς στο συγκεκριμένο θέμα. Πάντως καταλαβαίνετε ότι απαιτούνται επενδύσεις στο σύνολο του άξονα αυτού. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προσεγγίσουμε όλοι μαζί. Τα σενάρια δεν ε, είναι τόσο απεσιόδοξα όσο τα περιέγραψε ο κύριος Κράμερ. Ε, το 2043 θα έχει αναπτυχθεί το δίκτυο στην πληρότητά του. αλλά στο μεταξύ υπάρχουν άλλα μέτρα ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ε, ανάγκες. Ε, δεν ε, θα προσφύγουμε κατά των γειτονικών μας χωρών, συνομιλούμε μαζί τους. Και έτσι καταφέρουμε να πετύχουμε πρόοδο. Ο κύριος, Δεκα, ε, κύριος Φαντεκάμπ αναφέρθηκε στην χρηματοδότηση κατά τα δύο τρίτα ε, ναι, πράγματι, σε όλες τις χώρες νομίζω ότι είναι... Η ε, οι διεθνείς μεταφορές ε, χαμηλότερες από τις εγχώριες μεταφορές και έχουμε στην Ελβετία πολλά φορτηγά τα οποία προμηθεύουν τα εγχώρια καταστήματα. Εντός λοιπόν της Ελβετίας ε, έχει γίνει ε, συνεννόηση ε, μεταξύ των διαφόρων εταιριών μεταφορών και κάτι ακατανόητο για την Ευρώπη στην Ελβετία έχουμε συχνά μεταφορές αγαθών σε αποστάσεις 50-60 χιλιόμετρα. Ε, πάντως οι σιδηρόδρομοι αποτελούν ε, σαφές κομμάτι των ε, δικτύων μεταφορών εντός της Ελβετίας. Τα φορτηγά έχουν μια ειδική συσκευή, ακόμα και τα φορτηγά από το εξωτερικό συχνά έχουν τη σχετική συσκευή για πληρωμή των τελών χρήσιμο θα είναι κάποια στιγμή να έχουμε ενιαία συσκευή για το σύνολο της Ευρώπης. ο κύριος Έρτουκ αναφέρθηκε στην μείωση του θορύβου από το 2020 είπαμε πολύ συγκεκριμένα ότι δεν θα έχουμε σειρμούς που να παράγουν τόσο θόρυβο. Δεν πρόκειται για κάποια νέα δική μας εφεύρεση, απλά εφαρμόζουμε κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λίγο πιο αυστηρά. Είχαμε μεγάλες συζητήσεις, ο σχετικός κλάδος αντιστάθηκε σε κάποιο βαθμό αλλά βλέπουμε ότι αυξάνεται η κυκλοφορία σε αυτόν τον άξονα βορρά-νότου και πιστεύουμε ότι το 2020 θα έχουμε φτάσει σε αντακατάσταση των παλαιών σειρμών ε, σε ποσοστό σχεδόν 100%. Κάναμε λοιπόν τις σχετικές επενδύσεις επειδή ακριβώς θέλαμε να επιδείχουμε το στόχο αυτό. Αυτό συνδέεται όμως και με την αποδοχή από τους πολίτες. Ε, οι πολίτες μας ε, δεν θέλουν ε, μέσα μεταφοράς που να κάνουν τόσο θόρυβο. Μπορείτε να πετύχετε πολλά με τη δημιουργία κινήτρων, αλλά εάν ένας δεν συμμορφωθεί, τότε δεν κερδίζουμε τίποτα. Είχαμε λοιπόν προβλέψει μακρά μεταβατική περίοδο. Και θα χαρούμε πολύ αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον κάποιες χώρες μας ακολουθήσουν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, Όταν λάβαμε τη σχετική απόφαση, σκεφτήκαμε κάθε φορά στο τέλος του χρόνου να καθορίσουμε τι θα πληρωθεί την επόμενη χρονιά. Εάν λοιπόν η αρχή του υπολογισμού είναι το κοινοβούλιο, ε, δεν θα έχετε και επιλογή, διότι φαίνεται αυτομάτως πόσα ε, χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ειδικό ταμείο διότι μπορούμε ε, έτσι να κατευθύνουμε καλύτερα τις επενδύσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει δυνατότητα προσανατολισμού. Επίσης, στο σύνολο των σιδηροδρόμων έχουμε κατά νου ότι η υποδομή είναι κάτι πολύ γενικό. Δεν σκέφτεται λοιπόν κανείς ε, από τη μια χρονιά στην άλλη πως θέλουμε σιδηρόδρομο. Είναι κάτι το οποίο ε, γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εάν οι ανάγκες του τομέα είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα, τότε θα πρέπει ο Υπουργός ε, Μεταφορών να πάει στον Υπουργό Οικονομικών και να πει ότι θέλω περισσότερα χρήματα για τους ε, σιδηροδρόμους. Εάν επιχειρηματολογεί σωστά ε, θα λάβει τους επιπλέον πόρους, εάν όχι τότε απλά όχι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το ποια είναι η αρχή του προπολογισμού. Κύριε Κράμερ, επίση, ε, νομίζω ότι απάντησα όσον αφορά το 2020, όσον αφορά τα ποδήλατα στα τρένα. Τα τρένα μεγάλων αποστάσεων στην Ελβετία ε, επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων. Υπάρχει βαγόνι ειδικό. Αν δηλαδή δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτου στο τρένο ICE, πάρτε ελβετικό τρένο, εκεί μπορείτε. Επίσης, ακολουθούμε τις προδιαγραφές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν παρασχεθεί η υπηρεσία, ο επιβάτης μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματά του. Επίσης, όσον αφορά την αρχή του ρηπαίνοντος. Ε, με τις ε, κατηγορίες ε, του κατηγορίες οχημάτων ευρώ έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε το θέμα. Έχουμε για παράδειγμα την, τάξη, την κλάση Euro 6. Οι σχετικοί πόροι διατίθενται για τον συγκεκριμένο σκοπό. Δεν ε, εισραίουν δηλαδή οι πόροι από αυτά τα τέλη στον γενικό προϋπολογισμό. Έτσι με την πολιτική μπορεί κανείς να πετύχει διτό σκοπό. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας, ε, αλλιώς με στη διάθεσή σας. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελβετική ακρίβεια. Έχει μεγάλη σημασία βεβαίως να υπάρχουν έσοδα, αλλά να γίνεται και ε, χρηστή διαχείρισή τους. Εσείς έχετε μεγάλη, μακρά παράδοση ε, κύριε Φουγκλιστάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επίσκεψη που ελπίζουμε να μην είναι η τελευταία φυσικά. Θα συνεχίσουμε στις 2.30. Στις 2.30 θα τα ξαναπούμε εδώ. Γεια σας.